Yes, hello. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε σε αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ξεκινάμε με την ημερήσια διάταξη και την έγκρισή της. Την έχετε στους φακέλους σας και αν δεν υπάρχουν σχόλια εγκρίνατε. Χωρίς αλλαγές. Έχετε στη διάθεσή σας όλες τις γλώσσες πλήν της Ρουμανικής, όπως και τα πρακτικά της Δευτέρας Σεπτεμβρίου δεν που είναι στο φακελό σα. Και άρα εγκρίνονται και αυτά αν δεν προβληθούν παρατηρήσει. Έχουμε λοιπόν τώρα την εξασφάλιση και υψηλού ασφαλείας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση με συντάκτη την κυρία Πιλάρδα Καστήλιο. Πρόκειται για γνωμοδότηση. Έχουμε κάπου 14 λεπτά στη θέσή μας, 5 λεπτά η συντάκτρια, 2 ισχυοδησηγητές, 3 ε, ισχυοδησηγητές, 2 οι λοιποί συνάδελφοι και άλλα 3 λεπτά η Επιτροπή. Παρακαλώ να είστε αυστηροί στην τήρηση του χρόνου. Έχετε το λόγο κυρία Πιλάντζα Καστελιού. Ε, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με το νομοθετικό αυτό φάκελο που έχει να κάνει με το υψηλό επίπεδο ασφάλειας στα δίκτυα πληροφορικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως ε, συντάκτρια γνωμοδοτήσεως συγγνώμη, για την Επιτροπή μας, θα ήθελα να αναφέρω τα βασικά στοιχεία στα οποία εδράζεται η πρότασή μου, η οποία θα πρέπει να πάει στη μετάφραση στις 16 Οκτωβρίου. Μεθαύριο δηλαδή. Και όταν περάσει η διαδικασία της μετάφρασης θα έχω την ευκαιρία και πάλι να συναντήσω τους σκιώδους εισηγητέ. Για λόγους χρονοδιαγράμματος δεν μπορούσαμε να συναντηθούμε πριν από την 1η Νοεμβρίου, αλλά θα σας δώσω ε, ως ονούπο τη συγκεκριμένη ημερομηνία για τη συνάντησή μας. Είμαστε ενώπιον μιας πρότασης η οποία πρέπει να το υπενθυμίσω, ανταποκρίνεται στην αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2010 στην εκθεσή του για, μια ψηφιακή, για ένα ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και πιστεύω ότι είναι μια πρόταση η οποία είναι απαραίτητη γιατί αν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες που μας δίνει το ψηφιακό θεματολόγιο και οι οποίες ε, δυνατότητες αυτές έχουν να αντιμετωπίσουν το θέμα της ασφάλειας των δικτύων, κάτι το οποίο τώρα είναι πολύ επίκαιρο στα μέσα ενημέρωση. Έχουμε πάρα πολλές λοιπόν προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, οι οποίες απαιτούν μια κοινή εργασία από όλους μας, μια κοινή προσέγγιση, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληροφορικών δικτύων και είναι ακριβώς αυτό το αντικείμενο της πρότασης της Κομισιόν. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν πρέπει να αφήσουμε να περάσει αυτή η ευκαιρία, θα πρέπει να δείξουμε την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα και στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι το τέλος της ε, θητείας μας, ο οποίος είναι κάπως περιορισμένος, θα πρέπει να διεκπαιρεώσουμε το θέμα αυτό. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τώρα ποιοι είναι οι κύριοι άξονες ε, γύρω από τους οποίους θα πρέπει να αρθρωθεί η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πώς μπορούμε να συμβάλλουμε για να βελτιώσουμε την πρόταση της Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα, μια πρώτη βασική αρχή είναι η αρχή της αποτελεσματικότητας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί δεν θα πρέπει εμείς να περιπλέξουμε την ζωή μας αν αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν πρέπει να επισέλθουμε σε τομείς όπου δεν υπάρχουν περαιτέρω απαιτήσει οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν κάθε μορφή περί της γραφειοκρατίας και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας την ανάγκη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας. Επομένως, <clears throat> ακολουθώντας από την αρχή της αποτελεσματικότητας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, θα πρέπει να εξετάσουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Από την άποψη αυτή, η πρόταση της Κομισιόν, μέσω του παρατήματος υπαρτιμών 2, αναφέρει μια σειρά υποχρεώσεων που διευρύνουν τις υποχρεώσεις του κεφαλαίου 4 για σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Αλλά αυτός ο κατάλογος είναι κάπως ανοιχτός. Αυτό δημιουργεί προβλήματα. Προβλήματα γιατί παραμένουν ακόμα ασαφή ορισμένα στοιχεία αυτού του καταλόγου και επιπλέον προφανώς θα έχει νόημα να κρατήσουμε ανοιχτό αυτό το κατάλογο γιατί πάντα υπάρχουν νέα στοιχεία τα οποία μπορεί να προκύψουν και τα οποία θα πρέπει να μπορούμε να ε, ενσωματώσουμε αλλά το να είναι τόσο ευρύς ένας κατάλογος νομίζω ότι και αυτό μπορεί να είναι προβληματικό. Γιατί ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κουλτούρα ασφαλείας. Καλό είναι αυτό, αλλά συγχρόνως διατρέχουμε τον κίνδυνο <clears throat> να δημιουργήσουμε ένα πρόσθετο στρώμα γραφειοκρατίας σε ενωσιακό επίπεδο που θα είναι πολύ δύσκολο να, το, να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά οι κρατικές αρχές, παραδείγματο χάρη η αναφορά συμβάντων είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει δυσχέρειες στις ε, κρατικές αρχές και είναι απαραίτητο να έχουμε μια κουλτούρα κινδύνου που θα βασίζεται στην εκτίμηση κινδύνου και επομένω θα πρέπει να εμπλέκει σε διάλογο τους φορεί της αγοράς και τις αρμόδιες αρχές. Για μένα λοιπόν όλες αυτές οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 4 θα πρέπει να περιορίζονται μονάχα στις κέρυες υπηρεσίες, <clears throat> υπηρεσίες που έχουν κρίσιμο χαρακτήρα για την σωστή λειτουργία των ε, ψηφιακών υπηρεσιών, είτε είναι μεταφορές, είτε είναι ενέργεια, είτε είναι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Γι' αυτό πιστεύω πρέπει να τροποποιήσουμε σχετικά το παράτημα 2. Και για τις δημόσιες αρχές είναι απαραίτητο να εξεύρουμε μια ισορροπία μεταξύ των υποχρεώσεων που ήδη υπάρχουν για τις δημόσιες αρχές και την όθηση που θέλει να δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην, για να προωθηθεί η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στις δημόσιες αρχές. Πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη το ρόλο των δημοσίων αρχών, κάτι που προσπαθώ να κάνω και στην έκθεσή μου. Επίση, για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, είναι απαραίτητο να επανεξετάσουμε την πρόταση τη Κομισιόν για τη δημιουργία από κάθε κράτο μέλο μια αρμόδια αρχή, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση τη εφαρμογή αυτή τη οδηγία. Φυσικά, Υπάρχουν διαφορετικέ λύσει που μπορούν να ακολουθηθούν από τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτή τη οδηγία. Δεν ξεχνάμε ότι κάθε κράτος μέλος έχει τη δική του στρατηγική για ασφάλεια στον κυβερνόχωρο. Κάθε κράτος λοιπόν μπορεί να έχει την ανάγκη να θεσπίσει τομεακές αρχές ή αρχές που καλύπτουν ορισμένους μονάχα παρόχους κτλ. Αλλά το πιο λειτουργικό, το πιο σωστό δεν είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για νέες αρχές, να δημιουργήσουμε νέες αρχές, αλλά να έχουμε ένα ενιαίο σημείο επαφής μέσω του οποίου μπορούν να, να διοχετεύονται οι πληροφορίες. Να υπάρχει ένας λοιπόν εκπρόσωπος σε κάθε κράτος μέλος, ο οποίος να εμπλέκεται σε αυτό το δίκτυο συνεργασίας σε ενωσιακό επίπεδο και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν δημιουργήσουμε ένα άκαμπτο σχήμα μηχανισμών και αρχών σε κάθε κράτος μέλος, τότε θα πρέπει να δημιουργηθούν πρόσθετες αρχές και αυτό δεν είναι η καλύτερη λύση. Θα πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη ευκαμψία ώστε κάθε κράτος μέλος να χρησιμοποιήσει το μηχανισμό που επιλέγει, αλλά φυσικά να υπάρχει ένα ενιαίο σημείο για επαφές και συνεργασίες. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ομάδες άμεσης αντίδρασης σε συμβάντα ε, πληροφορικής, θέματα ασφάλειας, λεγόμενες SERT, θα πρέπει και αυτές να υπόκεινται σε αντίστοιχες ε, προδιαγραφές. Κάθε κράτος λοιπόν θα πρέπει να έχει τον τρόπο με τον οποίο θα δώσει το, την απάντηση σε αυτά τα συμβάντα με χρήση εθνικών, υποεθνικών, ιδιωτικών φορέων, ειδικευμένων ή γενικού χαρακτήρα, οριζοντίων ή μη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν τα διαφορετικά υποδείγματα τα οποία χωρούν στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση αυτού. αυτή. Και επίση η διακυβέρνηση τη κυβερνοασφάλεια σε κάθε κράτο μέλο. θα πρέπει να εναπόκειται στην επιλογή του κάθε κράτους μέλους, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι διάφορες σερτς, οι ομάδες άμεσης ε, αντίδρασης, θα πρέπει να σέβονται τις γενικές προδιαγραφές, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τις δράσεις προτεραιότητας επί τη βάση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυβερνοασφάλεια. Για μένα λοιπόν αυτή η οδηγία θα πρέπει να ζητήσει από τα κράτη-μέλη αποκλειστικά και μόνο ότι θα εξασφαλίσουν την ύπαρξη ομάδων ΣΕΡΤ οι οποίες θα μπορούν να λειτουργούν σε κάθε ένα από τους οικονομικούς τομείς που καλύπτονται από την οδηγία, από την οδηγία χωρίς όμως να επιβάλλει ένα συγκεκριμένο μοντέλο διακυβέρνησης σε κάθε κράτος μέλος. Δηλαδή να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη δυνατότητα συντονισμού για να υπάρξει διαλειτουργικότητα και δυνατότητα επαφής αλλά χωρίς να επιβάλλουμε ένα συγκεκριμένο υπόδειγμα να υπάρξει μια σειρά από ελάχιστες αρχές, ελάχιστες προδιαγραφές που είναι απαραίτητες για τον συντονισμό και τίποτα παραπάνω. Μια άλλη προτεραιότητα η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί ή καλύτερα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη στην πρόταση αυτή είναι η δημιουργία ενός κλίματος μεγαλύτερης εμπιστοσύνης τόσο για τους φορείς της αγοράς ώστε να μην φύγονται από την ανακοίνωση των συμβάντων στον κυβερνόχωρο και επίσης και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τις εθνικές αρχές για τους παρόχους υπηρεσιών, αλλά γενικά μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε όλους τους εμπλεκόμενους στο διαδίκτυο. Τελικά, ποιο είναι ο στόχο τη πρόταση, είναι να επιτύχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλεια στα πληροφορικά δίκτυα και δεν πρόκειται για μια οδηγία που αφορά τους καταναλωτές και γι' αυτό η δική μου πρόταση είναι, και θα παρουσιάσω τροπολογίες για το θέμα αυτό, για την ε, διατήρηση της εμπιστευτικότητας ορισμένων πληροφοριών. Πιστεύω ότι αυτό είναι απαραίτητο. Νομίζω ότι έχω ξεπεράσει τα πέντε λεφτά. Επειδή είναι περιορισμένο ο χρόνος μου, λοιπόν, θέλω τέλος να υπενθυμίσω ότι θα παρουσιάσω τροπολογίες σε σχέση και με τις κατά εξουσιοδότηση πράξεις και επίσης για, συγγνώμη, για την εφαρμογή που πρέπει να γίνει και τα, τις εγκυκλίες που πρέπει να αποστέλλονται στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή αυτή. Ε, αυτά, αυτή ήταν η σύντομη μου παρέμβαση. <coughs> Μεθαύριο θα στείλω στη μετάφραση την πρότασή μου και στις αρχές του Νοεμβρίου <clears throat> θα κάνουμε τις πρώτες επαφές των σκιωδών εισηγητών αφού έχουν όλοι στα χέρια τους τις μεταφράσεις και φυσικά παραμένω στην διάθεση όλων των ε, σκιωδών εισηγητών και των υπολείπων συναδέλφων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ε, εκπόνηση της γνωμοδότησής μας. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και νομίζω ότι όλοι μπορούν να συμβάλλουν για να εμπλουτίσουν αυτή την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Κλάντε, ο οποίος λαμβάνει τον, ε, το λόγο εξ του κύριου Χάλνταν για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και όντως θα σας διαβάσω τις ε, παρατηρήσεις του συναδέλφου γιατί δεν μπορεί να έρθει. Η στόχευση και οι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόταση για την εξασφάλιση κοινού επίπεδου ασφαλεία δικτύων και πληροφοριών θα πρέπει να διευρυνθεί. Βέβαια κάποια πράγματα ίσω να επαναλαμβάνουν τα λόγια τη κυρία Δεκαστήλιο αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ποια σημεία ή για ποιου λόγου θα πρέπει να κοινοποιείται μια παραβίαση, τι είδου υποχρεώσει έχουν οι αρχέ και πώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, έτσι ώστε να γίνεται σεβαστή και η ιδιωτικότητα και το απόρριτο και βέβαια να υπάρχουν διατυπώσει για, για τον τρόπο επικοινωνίας των αρμοδίων αρχών σε σχέση με την ε, πλατφόρμα ασφάλειας των δικτύων στην κοινοποίηση. Αν υπάρχει παραβίαση των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει αυτή να αντιμετωπίσετε με βάση τις νέες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου για την των προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να διευκρινιστεί σε με ποιο τρόπο τα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνονται παραγωγή υλικού και λογισμικού για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα πρέπει να αποκλείονται, αλλά θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία, θα πρέπει να διευρύνουμε τις προδιαγραφές ώστε να έχουμε ένα διατλαντικό επίπεδο. Η πρόταση του κυρίου Σφάπ από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς για την εξαίρεση από το δημόσιο τομέα του, των δημοσίων αρχών είναι απαράδεκτη. Η ασφάλεια της ανταλλαγής πληροφοριών δεν πρέπει να αποφασίζεται από τον ιδιοκτήτη του δικτύου, τον κύριο του δικτύου. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι ομάδες search, το, οι ομάδες δηλαδή επιβεβαίωσης ασφάλειας. Αυτές ήταν οι προτάσεις του κύριου Γκάλφιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλος ένας Γερμανός λοιπόν, ο κύριος Κρότσμαν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, το θέμα αυτό λοιπόν της ασφάλειας των δικτύων ε, προσλαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σημασία, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό ε, με επώδυνο τρόπο το αντελήφθημεν. θα πρέπει ιδιαίτερα να φροντίσουμε για τις όλο και αναπτυσσόμενες υποδομές και με μέλημα ιδιαίτερα τον καταναλωτή, γιατί αυτός αντιμετωπίζει προς τόσες συνέπειες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια καλύτερη συντονιστική προσπάθεια σε επίπεδο ευρωπαϊκό και να διευκολύνουμε τη δουλειά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Βασική η ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια σωστή ιδέα, αλλά σε αρκετά σημεία λεπτομεριών έχω κάποιες επιφυλάξεις προς το, πεδίο εφαρμογής. Είναι υπερβολικά ευρύ και δεν είναι ακόμη σαφέ ποιοι θα δραστηριοποιούνται. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφή όρια λοιπόν, ποιο θα είναι ο πάροχο, υπό ποιου ε, όρου θα ε, εντάσσει το σύστημα αυτό και ποιο όχι, τι είδου υπηρεσίε, ποιε θα είναι οι υπηρεσίε που πράγματι θα καταγράφονται. Ο τραπεζικό τομέα, ο τομέα τη ενέργεια, για παραδείγματι, έχει κεντρική σημασία τα δίκτυα και το online shopping, το ηλεκτρονικό εμπόριο θα περιλαμβάνονται ή όχι. Ε, γι' αυτό λοιπόν νομίζω πολλά ακόμα πρέπει να διευκρινιστούν και τίθεται το ερώτημα εάν, ε, ο, ε, εάν η πρόταση αυτή ε, επιτρέπει ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη και προστασία. Σε ορισμένους τομείς ήδη φύστανται συστήματα πάνω σε θελοντική βάση και δεν ξέρω αν υποχρεωτικό σύστημα θα αποτελεί βελτίωση κάποιοι τομείς μάλιστα οικονομικοί ξέρουμε ότι είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι και πιο προηγμένοι ως προς την ε, κυβερνοασφάλεια σχέση με κάποιους άλλους, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε μια ενιαία λύση και αντιμετώπιση και πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη και τις ε, ίδιες επιχειρήσεις και τα συμφέροντά τους, πράγμα το οποίο έχει να κάνει και με, τον, ε, με την εξυπηρέτηση του καταναλωτή αφενός, αλλά και με την προστασία του επαγγελματικού ή βιομηχανικού απορρίτου. Θα πρέπει ω εκ τούτου να εξασφαλίσουμε την προστασία των επιχειρήσεων από περαιτέρω επιθέσεις, ε, και η ροή των πληροφοριών θα πρέπει να βαίνει όχι μόνο, μόνο μερός, από πλευρά δηλαδή της, ε, της επιχείρησης προς ε, τις αρμόδιες αρχές, αλλά και αντίστοιχα, δηλαδή να υπάρχει το λεγόμενο feedback, αναφτροφοδότηση. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίσει η επιχείρηση σε ποια υπηρεσία θα πρέπει να στραφεί, ποια υπηρεσία εφαρμόζει ποιο μέρο τη διαδικασία, σε περίπτωση μάλιστα που δραστηριοποιείται σε διάφορα κράτη-μέλη μια, μια επιχείρηση και βέβαια στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι ακόμη πιο ασαφή. σω χρειάζεται μια εναρμόνιση, αυτό είναι μια λύση. Υπάρχουν λοιπόν κάποια σημεία ενδιαφέροντα μέσα στο κείμενο, δεν είμαι τόσο βέβαιο ότι αυτό μπορεί με την πρόταση τη συγκήτρια να αποτελέσει την ε, μοναδική λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κρότσμαν. Η κυρία Άντες Δότερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τον, την εισηγήτρια για την παρουσίασή της. Όπως τόνισε, είναι ένα σημαντικό θέμα και είναι πραγματικά κρίσιμο χαρακτήρα και είναι ένα δύσκολο θέμα για την ε, Επιτροπή μας. Υπάρχουν δύο μελέτες που τονίζουν ότι είναι ευρύ το πλαίσιο εφαρμογής αυτής της ε, Πρόταση και αρκετά μπερδεμένο. Εμεί θεωρούμε ότι το θέμα αυτό πρέπει να είναι ένα θέμα εσωτερική αγορά. Είναι σαφέ ότι το διαδίκτυο που χρησιμοποιούμε και για πολιτιστικό διάλογο, για ε, τραπεζικές ενέργειες, για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για καινοτομία, για ιδιωτικέ συνομιλίε, είναι ένα, ένας χώρος για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας χώρος όπου οι πολίτες και οι επιχειρηματίες μπορούν να οικοδομήσουν ένα καινούριο μέλλον. Είναι καλό το ίντερνετ για όλους μας. Η πρόταση τη Κομισιόν όμω έχει πολλά μειονεκτήματα και αυτό αναφέρθηκε και από του συναδέλφους μου. Αφενός, η κατεύθυνση τη πρόταση είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να κατανοήσω. Οι βιομηχανικοί κύκλοι είναι επικριτικοί, τα κράτη-μέλη φαίνεται ότι κατανοούν την κατεύθυνση αυτή τη πρόταση. Στη δική μου χώρα αυτή η πρόταση στάλθηκε στην Επιτροπή Άμυνα στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Από το πότε είναι η Επιτροπή Εθνική Άμυνα, ο χώρο για τον οποίο, στον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά πρέπει να πάει σε κάποια επιτροπή που ασχολείται με τα θέματα εσωτερική αγορά. Αλλά η δική μου χώρα μέλο δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι ήταν μια πρόταση που απευθυνόταν στα θέματα εσωτερική αγορά. Δεν είναι αυτό σκοπό η ασφάλεια. Είναι μέσο για να επιτευχθεί ένα στόχο. Θέλουμε η πλατφόρμα του ίντερνετ να είναι για όλου άξια εμπιστοσύνη. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε να υπάρχει όλο και μεγαλύτερη έλλειψη εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο, όπως φάνηκε και από τις ακροάσεις της ΛΥΜΠΕ για τα σκάνδαλα της NSA και της παρακολούθησης, τα προβλήματα που έχουμε να κάνουμε με το ανεπιθύμητο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και όλα αυτά. Η Κομισιόν το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να φτιάξει ένα χωριστό δίκτυο για τους σημαντικούς αξιωματούχους του, των κράτων μελών. Γιατί αυτοί λοιπόν πρέπει να έχουν ένα ειδικό δίκτυο και δεν πρέπει να υπάρχει ένα γενικό επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες πρέπει να παραμείνουν σε, ένα, σε μια πλατφόρμα που είναι το γενικό διαδίκτυο, όπου δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να είχε αντιμετωπίσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτή την οδηγία, αλλά βλέπω να υπάρχουν ελάχιστα βήματα προ το να γίνει κάτι για τον ευρύτερο κοινό και του πολίτε. Αυτό είναι λαθασμένο για μα. Ποιο θα ήταν ο λογικό τρόπο λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με μια οδηγία η ασφάλεια των δικτύων και της πληροφορίας στα κράτη-μέλη είναι κάτι που όλο και περισσότερο περνάει στα χέρια των στρατιωτικών φορέων. Οι ομάδες ΣΕΡΤ με τις οποίες έχουμε εργαστεί στην Επιτροπή μας περνάνε από, το τμήμα, από τα τμήματα βιομηχανίας και εσωτερικής αγοράς στους στρατιωτικούς. Δηλαδή οι στρατιωτικοί οι οποίοι είναι ακατάλληλοι για να αντιμετωπίσουν θέματα αγοράς ξαφνικά παίρνουν μια ευρεία ευθύνη για το πώ αντιμετωπίσουμε τα γενικά οικονομικά θέματα. Δεν είναι ένας φορέας ο οποίος καλλιεργεί την εμπιστοσύνη ο στρατιωτικός τομέας. Έχει μια ιεραρχική δομή. Εντάξει, αυτό είναι απαραίτητο για να αντιμετωπίσει κανείς στρατιωτικές ενέργειες και προβλήματα, αλλά θέλουμε μια πιο κατανεμημένη ευθύνη και μεγαλύτερη επικοινωνία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη στο γενικό επιχειρηματικό ε, χώρο που να βασίζεται και στην δημιουργικότητα και στην διάθεση συνεργασίας των ανθρώπων. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και διαφάνεια σε αυτή την οδηγία το ερώτημα είναι τώρα πώς μπορούμε να διορθώσουμε τα στοιχεία αυτής της ε, οδηγίας. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε σαφείς κανόνες για το ποιος έχει για οποιαδήποτε στραβοτημονιά την ευθύνη και συγκεκριμένα την αστική ευθύνη. Το να έχουμε στατιστικές είναι σημαντικό, αλλά οι στατιστικές που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ανύπαρκτες. Είπε η Κομισιόν ότι έχουμε κάπου από όλες 290 εκατομμύρια το χρόνο από κύβερνο έγκλημα, ενώ η, τα κέρδη είναι πολύ υψηλότερα. Δηλαδή κάποιος βγάζει 400 εκατομμύρια ευρώ, τη διαφορά ανάμεσα στα δύο, χωρίς να υπάρχει κάποιο τίμημα γι' αυτό. Η Κομισιόν έχει συλλέξει τα στοιχεία αυτά από εταιρείε οι οποίες δεν έχουν συγκρίσιμε στατιστικέ μεταξύ του. Πρέπει να ξέρουμε καλύτερα λοιπόν ποιε είναι οι απώλειε για να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη πολιτική για τα θέματα αυτά. Βλέπω ότι ετοιμάζεται να με χτυπήσει με το σφυρί ο πρόεδρο. Αλλά θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν πολλά σημεία σε αυτή την οδηγία όπου η Κομισιόν ξεκινάει σε μια καλή κατάσταση, σε μια καλή κατεύθυνση. Είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό σαν θέμα εσωτερικής αγοράς, αλλά κάποια προβλήματα που θέτει η Κομισιόν δεν δίνει λύση σε αυτά στην οδηγία και εμείς ως Κοινοβούλιο πρέπει να τα λύσουμε αν θέλουμε το διαδίκτυο να γίνει ομοχλός για μια νέα οικονομία όπως νομίζω ότι όλοι θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βίκη Φόρντ από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ και εγώ θα προσπαθήσω να σχολιάσω σε σχέση με αυτά που είπαν οι διάφοροι συνάδελφοι προηγουμένω. Ξεκινώντα με, με την συγκεντρία συντάκτρια, την οποία και ευχαριστώ ιδιαίτερω που επικεντρώνεται στου πιο σημαντικού τομεί. ενέργεια, μεταφορέ, υγεία, ματοπιστωτικές υπηρεσίε, όλα αυτά είναι πολύ σαφώ περιγεγραμμένα και ιδιαίτερω ευχαριστώ για την αναφορά στον σεβασμό των συστημάτων που ισχύουν σε ορισμένε χώρες, όταν είναι αρκετά αυστηρά ώστε να μην ε, ανατραπούν καλές πρακτικές. Πρέπει λοιπόν σε όλα τα κράτη-μέλη να υπάρχει το ελάχιστο επίπεδο της ασφάλειας των δικτύων και της κυβερνοασφάλειας μέσα από μια στρατηγική μέσα από ένα εθνικό σύστημα ομάδας ανταπόκρισης σε περίπτωση κινδύνου σχετικά με τα δίκτυα. Αμένα πλην όμως θα πρέπει να ε, μην ανατρέψουμε δομέ που λειτουργούν ικανοποιητικά στο ορισμένα Πολύ σωστά επισημαίνει τα συντάκτρια τα προβλήματα τη γραφειοκρατία, ειδικότερα για μικρότερε οργανώσει ή φορεί που ε, δεν γράφονται μέσα στους τέσσερις πρώτους ε, τομείς προτεραιότητας που μας περιέγραψε. Γι' αυτό λοιπόν καλό ήταν να γνωρίζουμε σαφώς ποιος τομέας, ποιος φορέας κάλυπτε από το πεδίο εφαρμογής της προτάσεως και επίσης τα σχόλιά σας για τις υποχρεώσεις του κλάδου Πιλάρ με βρίσκουν σύμφωνοι. Ελπίζω όμως και ο εισηγητής από την Επιτροπή Ιστορικών, Ιστορικής Αγοράς να ακολουθήσει αυτή την πρόταση και για τον ιδιωτικό τομέα αλλά και για το δημόσιο. Υπάρχει ανησυχία προς την αντιμετώπιση των απόρριτων πληροφοριών καλό θα είναι δηλαδή να μην είναι υποχρεωτική σε τέτοιο βαθμό η κοινοποίηση ώστε τελικά να κινδυνεύει η ε, εμπιστευτικότητα κάποιων πληροφοριών και τελικά να διστάζει κανείς να αποστελεί στοιχεία. Ε, διαφωνώ απολύτως με, τον, ε, με την πράσινη σκιώδη συγκεκριμένη η οποία από ό,τι βλέπω δεν έχει καν την αυροφροσύνη να ακούσει αυτά που έχουν να πούν οι συνάδελφοι, ούτε και ο πρόεδρος άλλωστο διαφωνώ, δεν έχει καμία σχέση με την άμυνα αυτό. Υπάρχουν στοιχεία ασφάλεια που έχουν τεράστιε επιπτώσεις προς την εθνική άμυνα και σε αυτό νομίζω θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη, όπως και τα θέματα της ιστορικής αγοράς, όσο και τα θέματα της ιστορικής αγοράς. Βεβαίως μπορεί να έχουν διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, κάποιες χώρες μέλη, αυτό είναι σημαντικό και για τις επιχειρήσεις. Βεβαίως η ελάχιστη εναρμόνιση είναι ε, η προοπτική αυτής της πρωτοβουλίας, γιατί μπορεί κάποιες χώρες να θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο στη νομοθετική του παρέμβαση και βεβαίως βλέπω ότι η συντάκτρια μιλάει για, το, ε, για την αρχή της εμπιστοσύνης για την εμφύσιση ε, εμπιστοσύνης σε αυτούς που ασχολούνται με το σύστημα, ώστε να φέρει πραγματικά αποτελέσματα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις επιχειρήσεις, ώστε να μην αποθαρρύνονται στη διάθεση πληροφοριών. Να λειτουργήσει λέει, το σύστημα με ε, παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς, ώστε να μην καθυστερεί και βρίσκεται πάντοτε ουραγός των εξελίξεων. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γόντε. Ε, μπορούμε να ακούσουμε τους ομιλητές, είναι ενδιαφέρουσες τροπολογίες. Έχετε δύο λεπτά. Πρώτος, το κατάλογο κύριος Τσουκαλάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναγνωρίζω τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε η Επιτροπή καταθέτοντας μια πρόταση για την κυβερνοασφάλεια που να είναι ασφα... αφενός αποτελεσματική και αφετέρου να είναι συμβατή με τις απαιτήσει των κρατών μελών και τις ιδιαίτερες ευαισθησίες που αυτά έχουν στο συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταλήγει σε συμβιβασμούς που καθιστούν την πρόταση αποσπασματική και εν τέλει αναποτελεσματική φοβούμαι ότι η τελική πρόταση περισσότερο εξυπηρετεί τι ανάγκης της γραφειοκρατίας της Επιτροπής, δηλαδή το να περιφρουρήσει ο κάθε επίτροπος από ένα πεδίο δραστηριοτήτων, cyber security, cyber crime, cyber war, παρά το να δημιουργήσει μια συνολική ευρωπαϊκή λύση που θα διασφαλίζει τα ασφαλή πληροφοριακά δίκτυα που οι κοινωνίες και οι οικονομίες μας έχουν ανάγκη. Το κείμενο καταλήγει στο να ακολουθεί κάποιες παραδοχές παραδείγματο χάρη για το που τελειώνει το cyber security και που αρχίζει το cyber crime ή για το που τελειώνει ένα εθνικό συμβάν cyber security και πότε αυτό κλιμακώνεται σε διεθνές ή παγκόσμιο, οι οποίες δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και με τα όσα συμβαίνουν στα δίκτυά μας, υποσκάπτοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ασφάλεια του διαδικτύου. Δημιουργούμε λοιπόν ένα πλαίσιο για την κυβερνοασφάλεια που εξυπηρετεί τους επιτρόπους και τα κάμπινετς, αλλά δεν είμαι βέβαιος σε ποιο βαθμό εξυπηρετεί την ασφάλεια για τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Βλέπουμε καθημερινά παραδείγματα του πώς επιθέσεις σε μεγάλες εταιρείες κλιμακώνονται μέσα σε δευτερόλεπτα και αποκτούν διεθνείς παγκόσμιες διαστάσεις. Μόλις τον τελευταίο μήνα είχαμε δύο μεγάλες κλίμακας επιθέσεις σε στόχους που θα περίμενε κανείς ότι γνωρίζουν καλά να προστατεύουν τους εαυτούς τους των οποίων είναι σαφές ότι το μέγεθος και οι επιπτώσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν με μεμονωμένες εθνικές υποθέσεις. Στην επίθεση της στη στη Γερμανία είχαμε απώλεια στοιχείων για 2 εκατομμύρια Γερμανούς πολίτες. Στην επίθεση στην Αμερικανική εταιρεία Adobe χάθηκαν τα στοιχεία 2,9 εκατομμυρίων πελατών μεταξύ τους και αρκετών Ευρωπαίων. Και κυρίως οι hackers απέκτησαν πρόσβαση στο πρωτότυπο προγραμματιστικό κώδικα που θα τις επιτρέπει τους επόμενους μήνες να πραγματοποιήσουν πολύ πιο στοχευμένες και μαζικές επιθέσεις. Φοβούμε ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι λύσεις που επιλέγει η Επιτροπή μπορεί να εξυπηρετούν την ίδια την Επιτροπή και να καλύπτουν τα ισχυρότερα κράτη-μέλη που έχουν ή νομίζουν ότι έχουν τους δικούς τους ισχυρότερους μηχανισμούς προστασίας του διαδικτύου. Όμως η ασφάλεια του πιο αδύναμου κρίκου ενός δικτύου είναι η ασφάλεια του υπολογιστικού συστήματος του ίδιου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τσουκάλα. Και για να ε, απαντήσω, η κυρία Άντερ Στότσερ με ρώτησε εάν μπορεί να απευθυνθεί στην Βρετανική αντιπροσωπεία για να κάνω μια ερώτηση. Ε, στη Βρετανική αντιπροσωπή λοιπόν, αλλά δεν μπορώ να σα δώσω το λόγο για να απευθυνθείτε. Α, και αν θέλει η κυρία Φόρτ προσωπικά να λάβει να δεχθεί ερώτηση από την κυρία Άντερ Στότερ, τότε εάν η κυρία Φόρτ το δέχεται, θα τη δώσω το λόγο τη κυρία Άντερ Στότερ, αλλά πρώτα η κυρία Φόρτ έχει να πείτε. Ναι, αλλά ξέρετε, η σκιώδη συγγήτρια από του Πρασίνου δεν με άκουγε. Εγώ του άκουσα όταν μίλησαν. Μετά σηκώθηκε Ήρθε να σας μιλήσει την ώρα που εγώ μιλούσα. Ε, δεν νομίζω ότι αυτό είναι ένδειξη σεβασμού ε, προς ε, συναδέλφους από μικρότερε ομάδε. Επομένω, δεν θέλετε να ακούσετε ερώτηση, λέει ο κύριος Ρόχοτε. Εάν είναι να μου ζητήσει συγγνώμη, να την ακούσω, βεβαίω. Μάλιστα, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, λέει ο κύριο Ρότε, αλλά πρώτα θα ακούσω τον κύριο Ηλή. Κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να επανέλθω στα όσα... Ο κύριος Έλερ να επανέλθω στα όσα υπόθηκαν. Ε, τώρα είναι διαφορετικές Το τοποθετήσεις, δεν μπορώ να πω ότι ε, συμφωνώ με τα όσα λέει η Επιτροπή κατά την κατανομή των αρμοδιοτήτων με την ΙΜΚΟ χάσαμε ό,τι αφορούσε τις σημαντικές παραγράφους. Ε, εμείς έχουμε μόνο γνωμοδότηση ενώ το διτακτικό το αποφασίζει η Επιτροπή των Ιστορικών Υποθέσεων. Γι' αυτό λοιπόν όταν θέλουμε να είμαστε σχετικά ε, φιλόδοξοι θα πρέπει να προσέχουμε και τι είδους αρμοδιότητες παίρνουμε και τι μπορούμε να γράψουμε μέσα σε ένα ε, κείμενο γνωμοδότησης. Έχει 130 περίπου τροπολογίες η Επιτροπή των, ε, της Εσωτερικής Αγοράς. Ξέρουμε ότι ε, το έβρος αυτό της συζήτησης εξαρτάται από τις οδηγίες που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών ε, προς τον ε, αρμόδιο εδώ πέρα. Αυτό ορίζει δηλαδή, το αντικείμενο της συζήτησης και αυτό που με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να πω ότι ε, οι συμβάσεις κινδυνεύουν αν δεν ρυθμιστεί το ζήτημα ικανοποιητικά και το έχουμε χάσει αυτόν τον αγώνα αρκετές φορές γιατί τα Υπουργεία, οι των Εσωτερικών μας λένε «Α, τις υποδομές για την ασφάλεια τις κανονίζουμε εμείς». Σε ένα ζήτημα έχει όμως δίκιο η συνάδελφος ότι εάν θέλουμε να κάνουμε έναν ορισμό ή ένα, να ορίσουμε ένα πλαίσιο ε, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τη συνθήκη θα πρέπει να ε, παραπέμπουμε στην εσωτερική αγορά και να μην μιλάμε μόνο για κρίσιμες υποδομές και ορισμούς αυτών. Γιατί εκεί δεν έχουμε αρμοδιότητα. Ως προς την εκούσια, την αυτοδέσμευση της, ε, του κλάδου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έτσι βιαστικά και γρήγορα αφήνουμε τους ε, επιχειρηματίες ε, της επιχειρήσεις να αυτοδεσμευτούν αν το θέλουν. Εδώ έχουμε να κάνουμε τεράστια συμφέροντα και προβλήματα και ανάγκη για προστασία του καταναλωτή. Γιατί λοιπόν ε, οι internet enablers, οι software και hardware producers και όλοι αυτοί να βγαίνουν έξω. Πώς θα ορίσουμε δηλαδή τελικά τις υποδομές. Και νομίζω ότι πρέπει με μεγάλη προσοχή να σκεφτούμε εάν πράγματι χρειάζεται ένα σύστημα αυτοδέσμευση, αλλά αν είναι έτσι τότε οι κλάδοι οι οποίοι είναι σχετικοί με την εσωτερική αγορά πρέπει να καλύπτονται και αντιστοίχω να δώσουμε και το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τους περιγράψει και να θεσπίσει τις διατάξεις που χρειάζονται. Αυτό όμως ε, δεν μπορεί να επιτρέψει ε, να περάσει η πρόταση της ΣΥΜΚΟ, η οποία ουσιαστικά ισοδυναμεί με την ε, λευκό επιταγή προς τις επιχειρηματίες, προς τις επιχειρήσεις. Εάν έχουμε να κάνουμε με, με εκούσια ρύθμιση, τότε θα πρέπει να διαβριθεί το αντικείμενο της αποκάλυψης στοιχείων, της δημοσιοποίησης. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με ε, παράλληλες εξελίξεις στη νομοθεσία σε άλλα κράτη, θα αναφερθώ στις ΗΠΑ σε παραδείγματα, ακριβώς το ίδιο αντικείμενο για, και αφορούν και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όπως και το, η δική μας νομοθεσία θα αφορά αμερικανικές, οι οποίες είναι πολύ πιο προχωρημένες από αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα λοιπόν ναι, θα πρέπει να προσδοριστεί η ε, ε, αυτοδέσμευση, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και αυτή η σχετική προσέγγιση για τους μετόχους. Πώς μπορεί δηλαδή μια αμερικανική επιχείρηση να υποχρεούται να αποκαλύψει τις απώλειες έσοδα λόγω της κυβερ... του κυβερνού εγκλήματος, σε παραδείγματα, και αυτό να μην συμβαίνει εδώ. Γιατί η κυρία Άντερ Στότερ μας λέει ότι ε, δεν θα πρέπει αυτό να καταγράφεται γιατί είναι ζημιέ, οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικό να καταγραφούνται στα λογιστικά βιβλία όταν προκαλούνται από το κυβερνό έγκλημα. Μα εδώ ακριβώς έχουμε να κάνουμε με ζητήματα στα οποία μπορούμε εμείς να συμβάλλουμε και αυτονόμως να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά στην ουσία της εκεί που μπορούμε να ε, προσφέρουμε μέγιστη υπηρεσία στην εσωτερική αγορά. Ιδάλλως παραμένουμε σε μια διακυβερνητική, διακρατική επαφή με πολύ περισμένε αρμοδιότητε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα επιτρέψω στην κυρία Σμόντι Ντότη να ε, θέσει ερώτημα, αλλά εξαρτάται από εσά αν θέλετε να απαντήσετε ή όχι. Ο λόγος που θα το επιτρέψω είναι γιατί ο κύριο με πλησίασε. Μάλλον κυρία Στόλτ με πλησίασε για να με ρωτήσει αν έχει το δικαίωμα να θέσει ερώτηση. Δεν ήρθε ω εδώ για να τα πούμε. Θα επιτρέψω λοιπόν να τεθεί το ερώτημα. Κυρία Στόλτ. Μα το ίδιο είναι, συνάδελφε. Δεν ακούσατε τη συνάδελφό μου και αυτό είναι το παράπονο. Μιλήσατε στον πρόεδρο. Είμαι βέβαιη, η κυρία Φόρντ θα με άκουγε. Είναι ικανή να κάνει δύο πράγματα παράλληλα. Θα ζητήσω συγγνώμη αν χρειαστεί. Παρακαλώ, ερώτησή σας να είναι σύντομη. Εάν απαντηθεί, θα δώσω το λόγο, εάν όχι, θα μείνει στον αέρα. Με συγχωρείτε, δεν ήθελα να υπάρξω αγενής. Η ερώτηση μου είναι, το Ηνωμένο Βασίλειο επενδύει 500 εκατομμύρια στερλίνες για να παρακολουθήσει μέσω του κυβερνοχώρου άλλα έθνη. Πώς μπορούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια κοινή αγορά να αισθάνονται εμπιστοσύνη για μια τέτοια πλατφόρμα και οι στρατιωτικές σας ε, δραστηριότητες, οι στρατιωτικές σας ενέργειες μας δημιουργούν καχυποψία. Έχουμε διαχωρίσει τα πράγματα αυτά για κάποιο λόγο. Το διαδίκτυο θα έπρεπε να χώρο για τους πολίτες, όχι για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πώς το εξηγείτε. you want to or... Θέλετε να απαντήσετε. Ωραία. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε τρία λεπτά. Κύριε Κάλγκορ. Ευχαριστώ. Κατά πρώτον, να ευχαριστήσω εδώ την Επιτροπή σας για την ευρεία στήριξη της πρότασής μας. Βεβαίως υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία χρήζουν διευκρινήσεων. Επιτρέψτε μου απλώς να θίξω τα πιο σημαντικά σημεία, διότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρώτα απ' όλα η εμπιστοσύνη είναι σαφώς ε, κέριο σημείο. Είναι μια από τις κινητήριες της οδηγίας αυτής, γι' αυτό και την προτείναμε, για να επικρατεί ένα κλίμα εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των ενδιαφορομένων και των κρατών μελών και εν ώψη της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Το πεδίο της οδηγίας προσπαθήσαμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί στηριζόμενοι στις υπάρχουσες δομές που λειτουργούν στι διάφορε χώρε χωρί να δημιουργούμε καινούργιε, για να υπάρχει ένα ελάχιστο κοινό επίπεδο ε, ασφάλειας ως προς, και πληροφορίε. ως προς τις πληροφορίες. Επίσης ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η κάλυψη των ε, φορέων της αγοράς που θα πρέπει να υπόκεινται στις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμερίζομαι τα σχόλια του κ. Έλλερ για τις κρίσιμες υποδομές εδώ η οδηγία θα έπρεπε να περάσει τα όρια των κρίσιμων υποδομών και να καλύπτει όλες τις βασικές εταιρείες διαδικτύου που λόγω ακριβώς της παρουσίας τους έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην δημιουργία της πολιτικής μας, της ψηφιακής ατζέντα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία ψηφιακή αγορά. Η παρουσία αυτών των υπηρεσιών είναι πολύ σημαντική για τη λειτουργία της κοινωνίας της πληροφορίας και της οικονομίας εν γέννη. Με την οδηγία αυτή θέλουμε βεβαίως να δημιουργήσουμε ίσους κανόνες του παιχνιδιού για όλες τις εταιρείε, που βεβαίως έρχονται αντιμέτωπε και με συνθήκες ανταγωνισμού. Πολλοί φορείς τηλεπικοινωνιών κάποιες φορές πρέπει να αναλάβουν ευθύνε που προκύπτουν από αυτή την οδηγία, άλλοι που θα εμφανιστούν σύντομα ή μπορεί να εμφανιστούν στο μέλλον, θα προτείνουν παρόμοιε υπηρεσίε, οπότε και αυτοί θα πρέπει να καλύπτονται για να υπάρχουν ακριβώς ίσοι κανόνες για όλους. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Κυρία Φόρντ, θέλετε το λόγο. Ναι. Να απαντήσω στην ερώτησή σας. Ήταν σαφής η παρατήρησή σας. Κατά την άποψή σας το θέμα αυτό είναι θέμα της εσωτερικής αγοράς και όχι θέμα άμυνας. Το καταλάβαμε. Αλλά όταν ε, ξαναπαίνετε το λόγο για να μου θέσετε ερώτηση, μέλους της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και ενέργεια για ένα θέμα αμυντική πολιτική του Ε.Β. που δεν είναι μέσα στι αρμοδιότητε αυτή τη Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Τι να σα πω. Την ερώτηση αυτή να τη θέσετε σε έναν εκπρόσωπο τη Βρετανική κυβέρνηση γραπτό. Θα βεβαιωθώ ότι θα φτάσει στα χέρια του υπεύθυνου Βρετανικού Υπουργείου και θα λάβετε απάντηση. Πιστεύω ότι υπάρχουν τμήματα του, του θέματος αυτού όπου μπορεί να υπάρξουν κενά και ελλείψεις στη λειτουργία του διαδικτύου. Ε, θέματα τεχνικά, ανθρώπινα σφάλματα, αλλά και κάποιες ε, κακόβουλες επιθέσεις. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν κακό να δούμε αυτά τα ενδεχόμενα σφάλματα που μπορεί να προκύψουν. Τώρα, για την ερώτησή σα περί αμυντική πολιτική, θα φροντίσω να προωθηθεί στου αρμόδιου για να δώσουν κάποια απάντηση. Εγώ όμω, στα πλαίσια τη Επιτροπή ε, Ενέργεια, Έρευνα και Βιομηχανία, δεν μπορώ να απαντήσω. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο λόγος τώρα στην εισηγήτρια για να ανακεφαλαιώσει. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν το λόγο. Σίγουρα μπορούμε να φανταστούμε ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις που θα ακολουθήσουν. Είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον και πάθος ακόμα. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το διαδίκτυο αφορά όλους, όλες τις ε, βιομηχανικές δραστηριότητε, αφορά τα άτομα, αφορά την ασφάλεια, αφορά το Βατικανό. Μιλάμε λοιπόν για το διαδίκτυο και στο βαθμό αυτό εξαρτάται από το τι βλέπει ο καθένας σαν προτεραιότητα μπορούμε να καλύψουμε όλα τα στοιχεία του επιστητού. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια πολυμορφία στο διαδίκτυο και αυτό ακριβώς του δίνει το μεγαλείο και τη σημασία και τον τεράστιο αντίκτυπο στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας στο γεγονός ότι υπάρχει το διαδίκτυο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο λοιπόν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το τονίσω περισσότερο. Νομίζω ότι αυτός ο πρώτος γύρος ε, παρατηρήσεων και έκθεσης απόψεων έχει παρουσιάσει πολλά στοιχεία με τα οποία εγώ μπορώ να ταυτίσω τον εαυτό μου και ήδη τα ανέφερα και προηγουμένως εγώ. Από αυτά που είπε ο κύριος Κάλφιν για το πώς πρέπει να γίνεται η, η ανακοίνωση των πληροφοριών μέχρι αυτόν που είπε η κυρία Φόρτ για το γεγονός ότι πρέπει να εστιάσουμε καλύτερα στο εύρος εφαρμογής αυτής της ε, πρότασης, τα ζητήματα ε, ανάγκη για αμφίδρομο διάλογο κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι μπορώ να συμφωνήσω με πάρα πολλά από αυτά που είπαν οι ομιλητές. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μπορέσουμε να εξετάσουμε ένα από τα ζητήματα τα οποία περιλαμβάνονται στην πρόταση της Κομισιόν που μπορούν να εμποδίσουν την συμμετοχή ε, ορισμένων στην ασφάλεια αυτή, παραδείγματος χάρη οι λίστες οι οποίες μπορεί να έχουν περιοριστικό χαρακτήρα και τονίζω και πάλι το γεγονός ότι πρέπει να είναι αμφίδρομος ο διάλογος, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και αυτές είναι ορισμένες πτυχές περιλαμβάνοντας τους καταλόγους που μπορούν να έχουν ένα κάπως τιμωρητικό χαρακτήρα για ορισμένου. Δεν πρέπει λοιπόν να αποκλείσουν από το διάλογο όλου αυτούς οι οποίοι θα πρέπει να είναι παρόντες και αντίθετα θα πρέπει να ενθαρρύνουμε το διάλογο. Πέραν όλων αυτών, εγώ θα προσπαθήσω να διαμορφώσω καλύτερα όλα αυτά τα οποία συμμερίζομαι από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια συγκροτημένη άποψη ως Επιτροπή Βιομηχανίας για το λόγο για τον οποίο πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο σε ορισμένα θέματα και αυτό μπορεί να αναφέρεται με πιο ε, εκτενή τρόπο στην αιτιολογική έκθεση. Αυτά λοιπόν και ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Νομίζω ότι θα υπάρχει και στο μέλλον τέτοια συνεργασία και πολύ έντονη μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κυρία Βελάρντ Καστίγιο. Να περάσουμε γρήγορα στην επόμενη έκθεση, έκθεση Περίρα. Μπαρέα, συγγνώμη. Έχουμε 40 λεπτά στην διάθεσή μας για αυτή τη συζήτηση. Διότι μετά πρέπει να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία στις 4 και 4. Να προσθέσω για το προηγούμενο θέμα ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι την 5η, ε, ε, λίγη την 5η 7 Νοεμβρίου. Κυρία Μπαρέα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση που αφορά κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές στην Επιτροπή μας και είναι αντικείμενο πολλών πρωτοβουλειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς δηλαδή θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ένα έφορο κλίμα για τις ε, επιχειρήσεις και ιδίως για τα λεγόμενα startups, για τις επιχειρήσεις που μόλις ξεκινάνε. Γι' αυτό είναι κάπως λιτή αυτή η γνωμοδότησή μου, αλλά θέλω να τονίσω περισσότερο το θέμα της πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσει η Ένωση για τις επιχειρήσεις, γιατί εδώ είναι ένα θέμα για το οποίο έχουν εγκριθεί πολλές οδηγίες, πολλές δράσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην πράξη δεν έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους λόγω της μη κοινή εφαρμογή ή τη εναρμονισμένη εφαρμογή κυρίω από τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία θέλω να τονίσω στη γνωμοδότηση αυτή είναι η ανάγκη να εναρμονίσουμε τη γραφειοκρατία, το θέμα των ευκαιριών που πρέπει να είναι ανοιχτέ σε όλου τα δίκτυα, το θέμα τη ε, ύπαρξη κεφαλαίου το οποίο θα πρέπει να επενδύεται και των χρηματοδοτικών εργαλείων, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσει είναι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση το πρόγραμμα κόσμε μας βρίσκει σύμφωνους, αλλά φοβόμαστε ότι είναι πάρα πολύ περιορισμένη η χρηματοδότησή του και επομένω κινδυνεύει να έχει ελάχιστο αντίκτυπο στι επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα COSME λοιπόν και το πρόγραμμα οι πολιετής δημοσιονομικές ε, προοπτικές έχουν κάποια χρήματα για την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της δημιουργίας απασχόλησης αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα όμως είναι να προωθήσουμε και το επιχειρήν και την κουλτούρα του επιχειρήν, της ανάληψης κινδύνου, ήδη στο σχολικό σύστημα, ήδη στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μελλοντικούς επιχειρηματίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε καλύτερες δυνατότητες δικτυακών πυλών που μας δίνουν μεγαλύτερη πρόσβαση και πληροφορίες για το δημόσιο εμπόριο, να έχουμε δημόσιες προμήθειε χωρίς εθνικούς φράκτες και επίσης να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει και κάποιος διάλογος μεταξύ των νέων επιχειρήσεων και των εδρεωμένων επιχειρήσεων σαν στοιχείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη των πρώτων. Θα καταθέσουμε και τροπολογίες για να συμπληρώσουμε αυτή τη γνωμοδότηση είναι περιορισμένο και ο αριθμό των λέξεων που μπορεί να περιλαμβάνει μια γνωμοδότηση όπω ξέρετε. Θα ήθελα λοιπόν να περιμένω τι τροπολογίε των συναδέλφων για τη βελτίωση αυτή τη γνωμοδότηση και ελπίζω να έχω τη συμβολή και όλων των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Κύριο Τσουκαλά. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισημάνω πω θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η έκθεση. Χρόνων ότι θα έπρεπε να έχει επιδείξει περισσότερη ε, δραστηριότητα προκαταβολικά η Επιτροπή μας και να έχει αναλάβει πρωτοβουλίες μέσω εκθέσεων που έχουν αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια και θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις μας και κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις να, καινοτομούν και να δημιουργούν τις θέσεις εργασίας που χρειάζονται σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της πληροφορίας. Καθώς βγαίνουμε λοιπόν ε, από την εποχή της κρίσης και βλέπουμε μια ανάπτυξη χωρίς θέσεις εργασίας και με 6 εκατομμύρια ανέργους στην Ευρωπαϊκή 60 εκατομμύρια μάλλον εννοεί ο ανέργους στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έρθει η στιγμή πλέον να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Πρέπει να δώσουμε κατεπίγουσα προσοχή στην υπόθεση αυτή, ιδιαίτερα για την πατρίδα μου. Παρά το γεγονός ότι έχουμε την πιο καλά καταρτισμένη γενιά νεαρών Ελλήνων αντιμετωπίζουμε ποσοστά ανεργίας 60% για τους νέους. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί είναι εκείνοι που φεύγουν στο εξωτερικό για να εργαστούν και έτσι υπονομεύεται η δυνατότητα της χώρας για ανάπτυξη για το μέλλον. Αυτό αφορά όμως όχι μόνο την Ελλάδα, είναι φαινόμενο που χαρακτηρίζει και άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οικογένειες και κράτη που έχουν επενδύσει πολύ μεγάλα ποσά για την κατάρτιση της νεολαίας τους, με, που τώρα έχει πτυχία παρεπιστημιακά, μεταπτυχιακά, ακόμη και δακτορικά και τώρα αναγκάζονται να μείνουν άνεργοι χωρίς να μπορούν να αξιοποιήσουν τα πτυχία τους, ε, τις γνώσεις τους και βρίσκοντας μόνο ε, κακοπληρωμένες δουλειές και αναγκάζονται να βρουν προσωρινές λύσεις μόνο. Ε, δεν υπάρχει δυνατότητα να βρουν λύσεις με δική τους ε, αυτόνομη επαγγελματική επιχειρηματική δραστηριότητα, περιορίζονται μόνο στις παραδοσιακές ε, μορφές απασχόλησης, ό,τι μπορούν να προσφέρουν οι επιχειρήσεις. Νομίζω ότι οι μικρές επιχειρήσεις που ξεκινούν θα δυσκολευτούν πολύ περισσότερο χωρίς τα μυαλά αυτά, τους άξιους αυτούς νέους που αναγκάζονται να φύγουν γιατί μόνο στην ε, Silicon Valley ξέρουμε ότι μπορούν να βρουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται. Η ψηφιακή οικονομία έχει τεράστιο δυναμικό δημιουργία θέσεων εργασία και ιδίω όταν σχετίζεται με του τομεί που παραδοσιακά έχει ισχυρή θέση η Ευρώπη, την ε, ε καινοτόμο τεχνολογία, τον τουρισμό, την, τον πολιτισμό ενώ στο παρελθόν χρειάζονταν περίπου 5 εκατομμύρια για να ξεκινήσει να παράγει ένα προϊόν μια νέα μικρή επιχείρηση, τώρα με τις νέες τεχνολογίες και τις ψηφιακές δυνατότητες προσφέρει το υπολογιστικό νέφος κτλ. έχει κόστος μόνο 30.000 ευρώ η αντίστοιχη δραστηριοποίηση νέας επιχείρησης. Άρα λοιπόν με προγράμματα όπως το Κόσμο Horizon και άλλα, μπορούμε να ενισχύσουμε επιχειρήσεις ε, να ξεκινήσουν ε, τη δραστηριοποίησή τους, όμως είναι πολύ περιορισμένη η χρηματοδότηση για αυτά τα ε, προγράμματα και δεν έχουμε περιθώριο. Πιστεύω να αφήσουμε να χαθούν αυτοί οι νέοι και να χαθούν οι ευκαιρίες για δημιουργία θέσεων και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων αυτών. Παρακαλώ. Είναι πολύ καλή η πρόταση γνωμοδότησης της κυρίας Άντρες Μπαρέα. Κάνει τη σωστή στόχευση και θεματοποίηση στο θέμα αυτό. Στην παράγραφο Γ αναφέρεται σε μία σειρά μέτρων αλλά εδώ πέρα έχουμε μονάχα το 2,5% του προϋπολογισμού της κόσμε. Εμείς θεωρούμε ότι το πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ακριβώς η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο θα δώσει σε αυτές τις επιχειρήσεις. Είναι φυσικά ε, ιδιαίτερα αξιέπαινη η πρόταση για μεγαλύτερο συντονισμό, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και στον τοπικό επίπεδο να υπάρχει η σωστή συνεργασία και να βρεθεί μια λύση ώστε το πολύπλοκο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θίγει το τοπικό επίπεδο. Είναι απαραίτητο επίσης να εξασφαλίσουμε και την συνεργασία των νέων επιχειρήσεων με τις εδρεωμένες επιχειρήσεις και αυτό πρέπει να ισχύσει ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες γιατί ακόμα έχουν πολλά προβλήματα για την πρόσβαση στην ψηφιακή αγορά και είναι δύσκολο να μπορέσουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε διαμεθοριακό επίπεδο και σε αυτό προστίθενται η πολυπλοκότητα της φορολογίας ΦΠΑ και δημιουργούν πραγματικά προσκόμματα στην ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ο κ. Λάμπερτς για τους Πρασίνους. Όχι, δεν θέλετε. Κυρία Φόρντ. Ευχαριστώ. Είναι ιδιαίτερα σημαντική έκθεση και αυτή. Λίγε μόνο παρατηρήσει. Αναφέρεται τη σημασία της, του περιορισμού τη γραφειοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφανώ συνεργάζεται με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει για να εντοπίσει ποιε είναι για αυτέ ε, οι δέκα πιο γραφειοκρατικώς επαχθείς νομοθετικέ πράξεις. Εμείς ως Επιτροπή όμως τι έχουμε κάνει για να μειώσουμε τη γραφειοκρατία σε αυτές τις πρώτες δέκα εκθέσεις. Θα πρέπει να αναφέρουμε συγκεκριμένε δράσει στο κείμενό μα για ακριβώ τα νομοθετικά αυτά τα οποία έχουν ε, πιέσει τι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως πλέον γραφειοκρατικές. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίε για να βελτιώσει την πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Αλλά πρέπει να κάνουμε και άλλα πολλά. Δηλαδή να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη όπου μπορούν να διευκολύνουν εκείνα τι μικρομεσαίε επιχειρήσει να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Και χρειάζεται περισσότερη τομεακή χρηματοδότηση πέραν από αυτή του δημόσιου τομέα. Όντω, ε, κάποιε χώρε φαίνεται να βρίσκουν το φω στην άκρη του τούνελ. Η Ιρλανδία, όπω άκουσα πρόσφατα στι ειδήσει, θα μπορούσε να ξεφύγει από την κρίση. Το Ηνωμένο Βασίλειο ε, ένα εκατομμύριο τέτοιες ε, θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν με 300.000 μικρομεσαίες startups τα τελευταία δύο χρόνια. Πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί τις υποσχέσεις της για την καλύτερη και ευφιέστερη νομοθεσία. Πρέπει να φροντίσουμε, να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία της νομοθεσίας σε περίπτωση που έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Ας δουλέψουμε λοιπόν καλά, ε, δίνοντας δυνατότητες και στην χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα πέραν του δημοσίου και ας μάθουμε από τα σφάλματα του παρελθόντος. Και ας δούμε κάποιες δράσεις επιτέλους, χειροπιαστές και συγκεκριμένε δράσεις. Ας αρχίσουμε να λέμε, να, να ονομάζουμε, τι, να δίνουμε όνομα σε αυτό που θέλουμε. Μια από τις ε, Δέκα οδηγίες λόγου χάρη είναι αυτή που αφορά το διαδίκτυο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποιες θα είναι οι ενέργειες που θα κάνουμε και πώς θα μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξεφύγουν από τις δυσβάσταχτες υποχρεώσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Βαρέα για το πολύ καλό αυτό σχέδιο γνωμοδότησης. Επισημαίνει κάποια σχόλια που είναι πολύ εύστοχα. Μιλάει για τον ουσιαστικό ρόλο του διαδικτύου, όχι μόνο για την διοργάνωση και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, αλλά και για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Επίσης τονίζει την ανάγκη τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν ε, εταιρικέ σχέσεις μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγαλύτερων εταιριών. Θα πρέπει να υπάρξει γεφύρωμα του χάσματος μεταξύ της ε, μόρφωσης και της ε, επαγγελματική ζωής και πολύ σωστά λέει ότι τα προγράμματα εταιρική σχέσης μπορεί να βοηθήσουν τις σχολές και τους φοιτητές που φοιτούν εκεί ώστε να σπουδάζουν μαθαίνοντας και βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους. Η Επιτροπή μα νομίζω σε αυτή τη γνωμοδότηση πρέπει να δώσει έμφαση στο ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση και να προωθήσουμε το πνεύμα του επιχειρήν και να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι οι δουλειές, οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται από τις επιχειρήσεις, όχι από την ε, ανάπτυξη του δημόσιου τομέα. Επίσης, να ακούσουμε προσεκτικά τις μέρημνες και ανησυχίες όσων είναι στο πιδάλιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και να θυμόμαστε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ευχαριστούμε ο κύριος Πρόντε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, διότι θεωρώ ότι είναι άκρος σημαντικό το θέμα, αλλά έγιναν ήδη κάποιοι σημαντικοί Πρώτα απ' όλα η πρόσβαση στα κονδύλια είναι το πλέον σημαντικό, χρηματοδότηση. Για όλες τις επιχειρήσεις, αλλά κατά κύριο λόγο για τις μικρομεσαίες. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται επίσης με τις γνώσεις για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και τη γνώση γενικότερα και να θυμίσω ότι ήταν πολύ χρήσιμες εδώ οι σχέσεις ιδιωτικού δημόσιου τομέα καθώς και οι συμπράξεις. οι κοινοπραξίες μάλλον για τη δημιουργία θέσεων εργασίας ε, είναι πολύ αποτελεσματικές ως προς τη δημιουργία υψηλότερου επίπεδου τεχνολογίας. Επίσης, ολοκληρώνοντας να τονίσω την ανάγκη να εμβαθύνουμε. Να εμβαθύνουμε στο σύστημα ανάληψης ευθύνης από τις υποχειρήσεις. Με την ε, social corporate responsibility όπως έχει ονομαστεί. Την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Θα πρέπει να διατηρήσουμε την απασχολήση σε ψηλά επίπεδα. Για να το πετύχουμε αυτό είναι ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε σημασία. Για να τονιστεί περισσότερο από το κέρδος και το εισόδημα αυτό το σκέλος και έτσι θα βοηθήσουμε στην πραγματικότητα της επιχειρήσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την ε, συνάδελφο, την κυρία Μπαρεά, διότι η πρόταση που επέβαλε είναι πραγματικά ιδιαίτερα έξυπνη για το πώς να δώσουμε μια όθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κάποιες ιδέες για το πώς να λειτουργήσουν καλύτερα και να αναπτυχθούν περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έκανε δυστυχώς όμως αυτό που έκαναν πολλοί άλλοι στο Ευρωκοινοβούλιο. Δηλαδή να επιδιώξω τη δημιουργία μιας τέτοιας θέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να βελτιώσουν τις θέσεις εργασίας ή το χρόνο εργασίας. Δεν είναι αυτός ο κατάλληλος δρόμος, η κατάλληλη τραπός. Ήδη στο πρώτο της σημείο η κυρία Μπαρέα τονίζει ότι υπάρχει κοινωνική ευθύνη. Αυτό τι σημαίνει. Ότι οι συλλογικές συμβάσεις για τις συνθήκες εργασίας και το καθεξής είναι μέρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό ε, θα πρέπει να θεωρείται τόσο θεμελιώδες δικαίωμα για κάποιον που δουλεύει σε μικρή επιχείρηση, όσο και κάποιον που δουλεύει σε μεγάλη. Υπήρξαν κάποιες εκθέσεις πρωτοβουλίας ως τώρα, οι οποίες ε, παρουσίαζαν και αυτήν την εκδοχή. Δηλαδή ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να αποτελούν εξαίρεση. Οπότε όσοι εργάζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μην διατρέχουν μεγαλύτερους κινδύνους από άλλους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Ουλσκοφ, ε, η Επιτροπή. Ο κύριος Ορμπέρ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Πολύ σύντομα για την βιομηχανική πολιτική ένα φιλόξενο περιβάλλον, ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Όταν μιλάμε για βιομηχανική πολιτική, τελικά τι καταλήγουμε να εννοούμε. Εννοούμε κάποιες συνθήκες πλαίσιο, ώστε να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να βελτιώσουν δηλαδή το δυναμικό τους και τις δεξιότητές τους και κατά αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε πλαγίως και τα προβλήματα της απασχόλησης και το καθεξής. Η πρόσφατη ανακοίνωση για την απασχόληση θέτει και σχεδιάζει προτείνει μάλλον τέσσερι πυλώνε που σχολιάζονται και στην έκθεση. Την πρόσβαση τη χρηματοδότηση και τι δεξιότητε. Αυτά ήταν τα δύο βασικά σημεία. Αυτό που κάνουμε τώρα στη φάση τη υλοποίηση, βέβαια, γιατί προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτέ τι πολιτικέ, είναι να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Όμω μεγάλο μέρο τη δουλειά τη υλοποίηση, είναι με εναρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σε μεγάλο βαθμό και των κρατών μελών και ιδίω των περιφερειών και των ε, ε, διαφόρων ε, αρχών τοπική αυτοδίκησης. Το συζητούμε λοιπόν στα αρμόδια φόρα για να δούμε πώ θα βελτιώσουμε την πρόσβαση στην χρηματοδότηση και να τονωθεί ταυτόχρονα η ανταγωνιστικότητα και η βιομηχανική ανάπτυξη. Να πω επίση ότι σε ομιλία του στι αντικαλιστικέ οργανώσει το Σεπτέμβριο, ο κ. Μπαρόζο τόνισε αυτή την διάσταση, λέγοντα ότι πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη βιομηχανική μα πολιτική. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και τώρα προετοιμαζόμενοι για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου. Εκεί θα συζητηθεί η βιομηχανική πολιτική. Συζητήθηκε και η γραφειοκρατία. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και το επιδιώκουμε εδώ και χρόνια να αντιμετωπιστεί με τη δουλειά μα για την καλύτερη νομοθεσία. Φέτο, όπω τα γνωρίζετε, ξεκινήσαμε κάποιου ελέγχου καλής υγείας, fitness checks όπως ονομάστηκαν για τις επιχειρήσεις, να δούμε τι προκύπτει από τις συνθήκες πλαίσιο και αν μπορούμε να τις βελτιώσουμε. Αυτό έγινε κατά κύριο λόγο στον τομέα των διηληστηρίων και του, της βιομηχανίας αλουμινίου. Εδώ κάνει λοιπόν ό,τι μπορεί με τις απαραίτητες πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Να δώσω και πάλι το λόγο στην κυρία Μπαρέα για να ανακεφαλαιώσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή τι ε, συνεισφορέ των συναδέλφων. Νομίζω όλε ε, οδεύουν προ την ίδια κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα, θεωρείται το σημείο αυτό ζωτική σημασία. Όντω, είναι σαν να διασχίζουμε την έρημο ε, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασία. Κάποιε χώρε έχουν μεγάλα προβλήματα με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενώ κάποιε άλλε είναι πολύ πιο προχωρημένες. Νομίζω όλα αυτά τα σχόλια που ακούστηκαν πάντως θα βελτιώσουν να εμπλουτιστεί η έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η προθεσμία για την υποβολή των απολογιών λίγη την Τρίτη στις 5 Νοεμβρίου το μεσημέρι, στι 12. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίε. Θα ξεκινήσουμε σε ένα δίλεπτο. Point of order, äh, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Μια παράκληση έχω. Ίσως θα είναι καλό για λόγους ε, χρονικούς να έχουμε όσο το δυνατόν τις ε, λεπτομέρειες των προγραμματιζομένων ψηφοφοριών. Μέχρι το Μάιο, α πούμε, να κάνουμε μια προβολή για να ξέρουμε τι μας περιμένει και να μπορούμε να οργανωθούμε καλύτερα. Ναι, λέει ο κύριος Ρόντε, αυτό σκοπεύαμε, αλλά εξαρτάται και από το πόση ώρα μιλάει ο κάθε συνάδελφος. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Από εκεί θα εξαρτηθεί το αν θα τηρήσουμε το πρόγραμμα. Ας περάσουμε όμως τις ψηφοφορίες. Πρώτα θα όμως θα κάνουμε τη δοκιμή του ηλεκτρονικού συστήματος. Άρχεται η ψηφοφορία. <laughs> That's not a good idea. <laughs> Vote is closed. The vote is closed. That's fine. Okay, we have a... Έχουμε ένα διαδικαστικό θέμα καταρχήν. Ναι, σας ακούω. Δεν έχετε την κάρτα σας. Εντάξει. Κυρία Ούλσκοκ, θέλετε το λόγο. θα ήθελα να ζητήσω να καταθέσω μια προφορική τροπολογία στην ε, συμβαστική τροπολογία 12. Το may να γίνει shall στα αγγλικά. Το δύναται να γίνει θα πρέπει να. Στο άρθρο 23 παράγραφος 1. Θα επανέλθουμε όταν φτάσουμε στο σημείο αυτό, λέει ο πρόεδρος. Εάν υπάρξει αντίρρηση από τέσσερα μέλη, τότε δεν θα γίνει δεκτή η πρότασή σα. Πρέπει να είναι τέσσερι οι οποίοι θα έχουν αντίρρηση. Τότε δεν μπορούμε να δεχτούμε, αλλά θα επανέλθουμε όταν φτάσουμε εκεί. Κυρία Άντερς Δότερ έχει επίσης διαδικαστικό θέμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όταν μπούμε στην ψηφοφορία θα ήθελα και εγώ να αναφέρω ότι δεν θα υποστηρίξει την ε, αυθεντικοποίηση στο διαδίκτυο αυτή η έκθεση και δεν πρόκειται να βοηθήσει την αγορά και τους παρόχους ε, υπηρεσιών, θα ξεπουλήσει ουσιαστικά την αγορά σε ξένα καρτέλ και παρόχους. Θέλω να προειδοποιήσω λοιπόν τους συναδέλφους για την τελική ψηφοφορία στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Έτοιμοι. Πάμε. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 111 μέχρι 114. 111, 12, 13 και 14 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 12 και 16 από κοινού είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνονται. 115 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1-16 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές δεκτή. 117 υπέρ κατά αποχές είναι κάπως ασαφές, τουλάχιστον για μένα. Ηλεκτρονικός έλεγχος είναι 117 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 20 με 21. Τροπολογία 118. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά. Από Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 129. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 Ιούρι. Θέλετε έλεγχο για την 128. Μάλιστα. Ηλεκτρονικός έλεγχο για την 128. Για την 129, συγγνώμη, 129. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 129. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται, 21-19. 130. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 λίμπε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 Γιώργη. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή 138 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 16. Θέλετε έλεγχο. 138 έλεγχος. Μάλιστα. Ελέγχουμε την 138. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 1326. Πάμε στη 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έλεγχος για την 159 λοιπόν. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 1.91 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτωτε 192 υπέρ. Κατά. Αποχές. Χρειαζόμαστε έλεγχο. Στην 192. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 193 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβεστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.27 και 71 από κοινού υπέρ κατά αποχές δεκτές. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 45 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 288 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 91 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 95 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 351 και 103 μαζί, υπέρ, κατά αποχές δεκτές. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Κύρια Ούλσκοφ, έχετε τώρα το λόγο. Θα ήθελα να έχω μια προφορική τροπολογία τώρα το πρώτο may θέλω να γίνει shall be. Αντί για may be, shall be. Στο άρθρο 23, παράγραφος 1. Ευχαριστώ. Αντιρρήσεις. Εντάξει. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ψηφίζουμε. Συμβαστική 12 με την προφορική τροποποίηση. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 74 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Σύμβαση 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 407 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 408 υπέρ κατά αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε 408. 408 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 409 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 410 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 411 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4-12 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για 412 παρακαλώ 412 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή 26-15 Συμβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 19. Υπέρ. <clears throat> Κατά. Αποχές. Δεκτή. 426. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν γίνεται δεκτή. Έλεγχος για 426. Μάλιστα. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 428 καθώς και 139 ταυτόσιμες άρχεται υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 429 θέλετε έλεγχο 428 και 139 βεβαίως η ψηφοφορία. 139. Πέρας. Εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. 429. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. Λέει ο μιλητής. Απορρίπτεται μάλλον. 20 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 434 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 434 άρχεται η ψηφοφορία πέρασε Εγκρίνεται. 435 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 συμβαστική υπέρ. Θέλετε να επαληθεύσουμε το 435. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 438. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 442 υπέρ, κατά, αποχές. Ε, απερίφθη. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 445 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Με συγχωρείτε, κάποιο λάθος κάναμε εδώ. Εγώ έκανα λάθος, λέει ο πρόεδρος. Γυρνώ στην 59 και 147 μαζί υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνονται. 447 ε, υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 448 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 449 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 54 υπέρ, κατά αποχές. Απερίφθη 55 υπέρ, κατά αποχές. Απερίφθη 56 υπέρ, κατά αποχές. Απερίφθη 59 υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται 61 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται θα έλεγα και επαληθεύουμε την 61 αρκετή ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 10 συμβαστική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 67 τροπολογία υπέρ, κατά αποχές. Κατά ε, απερίφθη. Υπαριθμόν 1 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη, 5 υπέρ, κατά χ εγκρίνεται 6 υπέρ κατά χ εγκρίνεται 22 συμβαστική υπέρ κατά χ εγκρίνεται 8 υπέρ κατά χ εγκρίνεται 5 υπέρ χ συγκρίνεται, εγκρίνεται συμβαστική 2α κατά χ εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά θα σηκώσετε τα χέρια σας καθαρά σας παρακαλώ υπέρ Ευρία πλειοψηφία εγκρίνεται. 73 τώρα παρακαλώ. Η τροπολογία 73 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη, παριθμόν 7 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη. 23 συμβαστική υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 75 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπάρχει μόνο 9 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 80 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 81 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 82 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 83 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά άποχες απερίφθη 89 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 90 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 μαζί με την 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 8 υπέρ κατά. Υπέρ παρακαλώ, στη χέρια. Κατά. Θα πρέπει να επαληθεύσουν. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τις ψηφοφορίες εγκρίνεται. Τροπολογία 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί. Και τώρα έχουμε μία τελική ψηφοφορία για τις τροπολογίες που υιοθετήθηκαν μαζί με το κείμενο, για το σύνολο του κειμένου, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τρία λεπτά υπέρ, 4 κατά, μία αποχή και ψηφίζουμε την πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τριαντεπτά υπέρ, τέσσερις κατά και εγκρίνεται. Vote on the interinstitutional negotiations and we need an absolute majority here. That means 30. Έχουμε λοιπόν 32 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 35 υπέρ, 4 κατά, 2 εποχές. Ναι, το ξέρω. Αλλά δεν είναι πρόβλημα. Έχετε την σας. Δεν πίεσα το κουμπί, δεν μετρήθηκε ψήφος μου. Συγχαρητήρια. The uh, Επόμενη ψηφοφορία της κυρίας Ντελ Καστιγιό για το cloud computing δίκτυο νέφους 33 τροπολογία 33 με την προφορική της τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, καταπίπτει. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, να ελέγξουμε για τον 28.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 Μπορούμε να αλλάξουμε την 33 αν θέλετε. Εντάξει, 34 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές καταπέπτει. 42 υπέρ κατά αποχές καταπέπτει. 43 δι υπέρ κατά αποχές καταπέπτει. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 και 51 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 52 υπέρ κατά αποχές αγκρίνεται 53 με την προφορική της τροποποίηση υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 54 θέλετε έλεγχο Ας ελέγξουμε. 53 με την προφορία και τη τροποποίηση. Άρχεται η προφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 και 61 υπέρ μαζί. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απολογία 1 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Ήμκο 1 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Ήμκο 2 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Ήμκο 3 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Ήμκο 5 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 3 υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. 13 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λίμπε 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λίμπε 4 μέρος 2 υπέρ, κατά, αποχές, καταβήτη. Λίμπε 6, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λίμπε 9, τμήμα 1, υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνουν. Ε, καταπίπτει. 13. 14 μάλλον. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λίμπε 26. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28. Μήμα 2. Υπέρ, κατά, αποχές, καταπίτη. 2. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9, 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άλτη ψηφοφορία. Πέρας. 41. Μία αποχή Συγχαρητήρια. Περνάμε στην επόμενη έκθεση, Σαρτόρη, για την ε, Ευρωπαϊκή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό GNSS. 47 υπέρ. Με συγχωρείτε. 47 υπέρ. Κατά. αποθέσεις απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 και 49 μαζί. Είναι πανομοιότυπες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές θα ήθελα να το ελέγξουμε. 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. Απορρίπτεται μάλλον. 15 προς 24. Περνάμε στην έκτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 και 10. Μαζί. Κατά. Αποχές δεκτές. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 53 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτονται. 54 και 57 μαζί. Υπέρ κατά αποχές ε, δεκτές. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 55 και 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 και 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. τεκτές Έλεγχος του προϋπολογισμού 1. Υπέρ. Κατά. Δεν βλέπω χέρια. Πάλι. Κοντ 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Κοντ 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5. 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 59 υπέρ με προφορική τροποποίηση του εισηγητού υπέρ κατά τις εισηγητές. Κατά δεκτή. 60 υπέρ με τροποποίηση υπέρ κατά αποχές δεκτή. 61 με τρο... προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 52 εκπίπτει, πάμε στην 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Κοντ 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 25 και 40 υπέρ κατά αποχές δεκτές. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 28 υπέρ κατά αποχές Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 66 υπέρ <clears throat> κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 67 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 31 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 34 <clears throat> υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 35 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή κοντ 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 37 και 38 μαζί υπέρ κατά κατά αποχές δεκτή κοντ 6 ναι εκπίπτει πάμε στην 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή 41 και 15 υπέρ κατά αποχές δεκτές κοντεπτά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42, 43 και 44 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κοντ 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ, κατά, υπέρ μάλλον, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, τρία, υπέρ, κατά, αποχές. Η 45 εκτύπτει διότι ενεκρίθη η 4. 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται εγκρίνεται, συγγνώμη λέει διορθώνει πρόεδρος, 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως έχει τροποποιηθεί η έκθεση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 38-0 με μία αποχή. Εγκρίνεται. Έχουμε τέσσερις τροπολογίες για το νομοθετικό ψήφισμα από την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Το νομοθετικό ψήφισμα όπως έχει τροποποιηθεί Ηλεκτρονικά, παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 39-0 με μία αποχή. Και τώρα η εντολή για τις <clears throat> διαθεσμικές διαπραγματεύσεις. Χρειαζόμαστε από την πλειοψηφία εδώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 39-0 με μία αποχή. Εντάξει. Συγχαρητήρια στην κυρία Σαρτόρη. Τέρμα η ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας. Να περάσουμε τώρα στο πρόγραμμα Κοπέρνικους. να δώσω στους συναδέλφους ένα λεπτό για να φύγουν από την αίθουσα. If you feel like discussing the votes, please... Εάν θέλετε να συζητήσετε τα αποτελέσματα των ψηφοριών, παρακαλώ εκτός αιθούσης, διότι ακόμη έχουμε κάποια χρονική πίεση Okay, we can start the discussion. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το πρόγραμμα Κοπέρνικους. Απευθείας να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας. Στην εισηγητρία μας από την κυρία Ρασίντα Ντατή. Όχι, όχι κύριε Πρόντι, με συγχωρείτε. Κύριε Πρόντι, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, εσείς είστε εισηγητής. Μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντατή. Κύριε Πρόντι, έχετε το λόγο, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινώ με την εισαγωγική παρατήρηση ότι ο κανονισμός ε, για το Κοπέρνικους, το οποίο αναμένουμε από καιρό, έφτασε επιτέλους μπροστά μας μετά από κάποια κόποση της όλης διαδικασίας. Κυρίως γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έπρεπε να περιμένει τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και να ετοιμάσει τον προπολογισμό για το Horizon 2020 και για το Γαλιλαίο πριν περάσει στην εξέταση του Κοπέρνικους και σε ό,τι απομένει να διευθετηθεί και να χρηματοδοτηθεί στην πολιτική του διαστήματος. Προκύπτουν ε, δεδομένα ε, χρονικά και τεχνικές δυσκολίες ώστε να καθιστούν το θέμα αυτό ιδιαίτερα κατεπήγον. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εξέταση πριν τελειώσει η θητεία του Ευρωκοινοβουλίου. Και έτσι ολόκληρο το πρόγραμμα και ο κόσμος ε, καθώς και εργαζόμενοι που από το πρόγραμμα αυτό, περιμένουν με ανυπομονησία για να αποφύγουν αρνητικές ε, συνέπειες. Κάποιε δραστηριότητε θα μπορούσαν να ακυρωθούν, να ανασταλούν εφόσον δεν υπάρξει ο τήσο προπολογισμό εγκαίρω. Δεν μπορούμε να περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρώσει τον κύκλο τη γραφειοκρατία, γιατί υπάρχουν και κάποιε προθεσμίε τεχνικέ ή τεχνολογικέ που καθορίζουν για παράδειγμα τη διάρκεια ή τη λειτουργία ενό δορυφόρου. Σε τέτοιους καιρούς κρίσης, η καθυστέρηση στην δημοσιοποίηση του κανονισμού θα επιδεινώσει μια κατάσταση που ήδη σε τετοιου καιρου κριση η καθυστερηση στην δημοσιοποιηση του δύσκολη. Ε, Κάνω έκκληση λοιπόν προς όλους τους συναδέλφους να κατανοήσουν ότι υπάρχει αυτός ο κατεπήγων χαρακτήρας και να αναζητήσουμε από κοινού ενδεχόμενες λύσεις για να αντιμετωπίσουμε διαφωνίες ή τέλος πάντων ε, διαφορετικούς προσανατολισμούς. Βεβαίως δεν θα πρέπει να θυσιάσουμε το τόσο καλό έργο που έχουμε πραγματοποιήσει στον τομέα του διαστήματος, ο οποίος είναι στατηγικός τόσο για την μηχανική ανάπτυξη της Ευρώπης όσο και για την ασφάλεια και την προστασία της επικράτειας της Ευρώπης και των πολιτών. Κάτι που θέλω να προσθέσω για το μέλλον του προγράμματος αυτού ε, έχει να κάνει με την οικονομική διάσταση. Θυμίζουμε ότι η μάχη που ξεκίνησα ε, προασπιζόμενο στο GMES στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και μάλλον του στόχο είχε να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης όπως και ίσχυε και στον προηγούμενο κανονισμό. Μετά από αμέτρητες ε, διαβεβαιώσεις του Συμβουλίου και κάποιων συναδέλφων του Ευρωκοινοβουλίου ανακαλύψαμε ότι αντιθέτως το Κοπέρνικους μπορεί να στηρίζεται μόνο σε έναν μειωμένο προπολογισμό 35-37% διατηρώντας ωστόσο τις ίδιες ευθύνες που προβλέπονταν ε, σε σχέση με έναν πλήρη προπολογισμό. Εάν το πρόγραμμα τελικά ε, μείνει ως είχε και έτσι ε, υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώ και δεν ακούστηκε καθένα αρνητικό σχόλιο από το Συμβούλιο εκείνο το διάστημα. Αν παραμένει λοιπόν μια προτεραιότητα για την Ένωση και εδώ συμφωνώ τελείω ότι για τι πολιτικέ του περιβάλλοντο, τη βιομηχανία, των κλιματικών αλλαγών, τη γεωργία, τη υγεία, τη ασφάλεια και ούτω καθεξή. Εάν λοιπόν παραμένει μια προτεραιότητα, έλεγα, δεν μπορούμε κάθε φορά να συνεχίσουμε να αμφισβητούμε επενδύσει που θα πρέπει να διατηρήσουν μια σχετική σταθερότητα για τουλάχιστον 15-20 χρόνια προκειμένου να μπορέσει να αποδώσει καρπούς σε επίπεδο της αγοράς αυτό το πρόγραμμα και για να υπάρξει συνοχή και επιστημονική αλλά και ανταγωνιστικότητα. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να ε, ολοκληρώσουμε την εξέταση εγκαίρως πριν από την εκπνοή του προηγούμενου κανονισμού και αυτό σε ένα πλαίσιο διαφοροποιημένης χρηματοδότησης που να είναι σταθερότερη, πιο μακροπρόθεσμη και που να προβλέπει διαφορετική διάρθρωση στις σχέσεις των διαφόρων φορέων. Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν παρουσιάζει μεγάλες εκπλήξεις σε σχέση με τον προηγούμενο, καθώς ε, το πρόγραμμα ονομαζόταν ακόμη GMES. συνολική παρακολούθηση για το περιβάλλον και την ασφάλεια. Στην έκθεσή μου όμως προσπαθώ να διοργανώσω την προηγούμενη δομή, ε, προσεγγίζοντας την περισσότερο στον κανονισμό GMES, ε, προσθέτοντας κάποιες προτάσεις για τις δημόσιες προμήθειες, ε, διατάξει τι οποίε αντέγραψαν απευθεία από τον κανονισμό για τον Γαλιλαίο και όπω είχαν συμφωνηθεί στους τριμερείς διαλόγους μεταξύ των θεσμικών οργάνων, αλλά και τον ρόλο του στην στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το Διάστημα. Στην πραγματικότητα, κατά την άποψή μου, τα δύο ζωτικά σημεία του κανονισμού είναι η πολιτική των δεδομένων και η governance, η διακυβέρνηση. Είμαι πεπισμένο ότι αυτό το πρόγραμμα, ω κοινοτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με τα κονδύλια, τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών, όταν θα αποφασίσουμε πώς να τα επενδύσουμε τα χρήματα αυτά, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τον έλεγχο για τις δαπάνες και τις ευθύνες που προκύπτουν από αυτές, όλες αυτές θα πρέπει να παραμένουν στο πλαίσιο της ε, ε, δημόσιας λογοδοσίας. Ως προς το ρόλο και την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού του Διαστήματος, αναφέρω ως προς τον κανονισμό στοιχεία που ήταν γνωστά και από το GMES ε, και προσαρμόζοντα τι διάφορε αρμοδιότητε στην φάση ανάπτυξη του προγράμματο. Σε σχέση με τα δεδομένα, δεν υπάρχει κάτι να προσθέσουμε πέραν το ότι θα πρέπει να μην υποχρεώσουμε του πολίτε να πληρώσουν για δεύτερη φορά για δεδομένα των οποίων η παραγωγή είναι κάτι στο οποίο έχουν ήδη συνεισφέρει. Η πλήρη πρόσβαση και ο δωρεάν ε, χαρακτήρα είναι κάτι που θα πρέπει να παραμείνει ενδιαφυσβήτητο. Σε ό,τι αφορά τώρα την ανταγωνιστικότητα, εάν χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να έχουν πρόσβαση ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα που είναι η βάση για τι δραστηριότητε πολλών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στι διεθνεί αγορέ, αυτό πρέπει να συζητηθεί. Πιστεύω ότι η πρότασή μου να διασφαλίσει τουλάχιστον την, την αμοιβαιότητα στι ανταλλαγέ δεδομένων με τρίτε χώρε είναι μια πιθανή λύση. Αλλά είμαι διαθέσιμο να τη συζητήσω και να τη βελτιώσω. Θα πρέπει έπειτα να αναζητήσουμε μια συμβαστική λύση για το πώ θα πρέπει να διοργανωθεί το Κοπέρνικου και το Κοπέρνικου Κομίτη, Επιτροπή για το Κοπέρνικου. Δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να δημιουργήσουμε έναν εσωτερικό κρίκο όπω ονομάζεται και το Core Users Forum ή κάποιον άλλο λιγότερο σημαντικό χωρίς δυνατότητες να λαμβάνει αποφάσεις. Γι' αυτό ένα δίκτυο που να αφοσιωθεί στην διανομή των δεδομένων, όπως είχε προταθεί και στην Ένωση των Περιοχών Νηρέας, αυτό θεωρώ ότι είναι το ιδανικό εργαλείο για να μπορέσουν οι πολίτες και οι πραγματικοί τελικοί χρήστες να έχουν στα χέρια τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το χρήση του Κοπέρνικους. Ε, στο κάτω-κάτω της γραφής, η πρόθεση όλη αυτή της προσπάθειας είναι να περάσει από τη φάση του σχεδιασμού στην αξιοποιήσει των υψηλότατων δυνατοτήτων του προγράμματο για να δημιουργήσει μια ad hoc αγορά. Ολοκληρώνοντα, να επαναλάβω ότι είμαι ανοιχτό σε επικοδομητικέ προτάσει και ευχαρίστω θα ακούσω τι απόψει των συναδέλφων που πάντοτε θεωρώ εξαιρετικά πολύτιμε. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Thank Ευχαριστούμε πολύ, κυρία. Και τώρα. Παρακαλώ την κυρία Γασίντα Ντατή να Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόντι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θέλω καταρχάς να συγχαρώ τον κύριο Πρόντι για την εξαιρετική δουλειά που έκανε στην έκθεση αυτή και να του ε, επισημάνω ότι συμφωνώ απολύτως μαζί του στο σύνολο των προτάσεών του και κυρίως προς την ανάγκη της επαγρύπνησης όσον αφορά την χρηματοδότηση κυρίως. Τα σημεία στα οποία παίζει δυσκολίε, είναι πραγματικά προβλήματα και πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Ιδιαίτερα δεν θα πρέπει να εμφαθύνουμε στο ρόλο των μεν και των δε, ώστε να είναι σαφής και ως προς τη στάση στο πρόγραμμα Κοπέρνικου, το πεδίο εφαρμογής και τους ορισμούς. Ναι, διευκρινίζει ο στο ρόλο της Επιτροπής και το καθεστώς των δημοσίων αγορών. Αυτό είναι θετικό. Για τους δίκτες προτείνει βελτιώσεις ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και χρήσιμοι. Ο ορισμός άλλωστε των δικτών αυτός είναι. Ε, ένα δείκτης θα πρέπει εξ ορισμού να είναι χρήσιμος και αποτελεσματικός. Για, τους, ε, για τις σκέψεις πρέπει να είναι βέβαια φορέας ανάπτυξη ένα τέτοιο πρόγραμμα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσεως, όσον αφορά το ρόλο του κλάδου. Ε, χαίρομαι για την σημασία, την αυξημένη σημασία που του δίνουν οι συγητής ως προς την ε, θέση εφαρμογή του προγράμματος, κάτι το οποίο έλειπε από τις προτάσεις της Επιτροπής. Μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι η Επιτροπή λησμονεί το ρόλο του κλάδου, της βιομηχανίας, του παραγωγικού κλάδου, ε, στην ανάπτυξη στην Ευρώπη. Μπορούμε να παραμείνουμε λοιπόν στις γραμμές που μας προτείνει ο εισηγητής, με, με κάποιες μικρές τροπολογίες στο ίδιο μήκο Για την αεροναυπηγητή εκεί βεβαίως θα έχει πολύ μεγάλη σημασία, ώστε το Κοπέρνικους να μπορέσει να αναπτύξει πλήρως το φάσμα των δυνατοτήτων του. Αμοιβαιότητα, συμφωνούμε με τον εισηγητή. Δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανεί την προσέγγιση που υιοθετεί. Τα δεδομένα δηλαδή θα πρέπει να ε, ανταλλάσσονται με εταίρου εφόσον αυτοί μα ε, επιτρέπουν την πρόσβαση στα δικά του δεδομένα, αλλιώ δεν έχει νόημα. Και ως προς την ε, πλαισίωση της έννοιας της αμοιβαιότητας πρέπει να είναι σαφής ο ορισμός της για να μην έχουμε προβλήματα εφαρμογής και ερμηνείας ώστε να, μην, έχουμε όρους ισότιμου ανταγωνισμού, ισορροπημένου ανταγωνισμού κτλ. Δεν θέλουμε η Ευρώπη να διαθέτει δωρεάν τα στοιχεία της στον πρώτο τυχόντα. Ήρθε η στιγμή να επιμείνουμε στην αυτών των δεδομένων και χαίρομαι για την πρόταση να παραμείνουν ανεκτά και ε, προσβάσιμα δωρεάν τα δεδομένα σε περίπτωση ενίσχυση της ανάπτυξη. Ε, η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, βλέπουμε να τροποποιεί το ρόλο της αεροναυπηγικής ε, και της σχετικής υπηρεσίας χωρίς να εξηγεί την επιλογή αυτή αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επανέλθω προς τις επικρίσεις μου προς το ρόλο της Επιτροπής σχέση με κάποια πράγματα κάπως παράδοξα που μπορεί να μας προτείνει. πέραν αυτού λοιπόν μπορεί και άλλοι φορείς, παράγοντες, δημόσιοι ιδιωτικοί να ε, είναι χρήσιμη για την ανάπτυξη του ρόλου αυτού πέραν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλωστε και εμείς δεν θα πρέπει πιστεύω να απεκδηθούμε των αρμοδιοτήτων και ευθυνών μα σε σχέση με την υπηρεσία του διαστήματος. Πρέπει με κάποιο τρόπο να την πλησιώσουμε ή να την ελέγχουμε εμείς ως κοινοβούλιο, γιατί δεν νομίζω ότι βλάπτει δημοκρατικός έλεγχος στις δράσεις που αναπτύσσονται κατόπιν εντολών και εκτελέστικών αρμοδιτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύ καλή η επιλογή του, του συντάκτη επομένω, απλώς θέλω να είμαστε λίγο πιο απαιτητικοί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντατή. Και τώρα θα πρέπει να λάβω εγώ το λόγο. Γιατί είμαι και εγώ σκιώδης συγητή για τους φιλελεύθερους. Η ομάδα μου χαιρετίζει την πρόταση της Κομισιόν σε σχέση με το πρόγραμμα Κοπέρνικος και θα ήθελα να πω επίσης ότι συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπε η κυρία Ντάτη. Και επίσης θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή μας τον κύριο Φρόντι για το ιδιαίτερα αφοσιωμένο έργο που έχει φέρει σε πέραση για το θέμα αυτό. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Απλώς θέλω να υπογραμμίσω ότι χαίρομαι πάρα πολύ να δω ότι προτείνει ο κύριος Πρόντι να υπάρξουν περιορισμοί σε σχέση με την πρόσβαση, την δωρεάν πρόσβαση για το πρόγραμμα αυτό σε χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τον Κοπέρνικο επί τη βάση της αρχής της Χαίρομαι επίσης που ο εισηγητής πρότεινε να υπάρξουν δίκτυα, ένα δίκτυο για τη διανομή δεδομένων που εξασφαλίζει την πρόσβαση στα δεδομένα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους εθνικούς φορείς. Κάτι όμως το οποίο θέλω να πω έχει να κάνει με την οργάνωση του προγράμματος. Η πρόταση της Κομισιόν λέει ότι η ΕΣΑ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, δεν θα έχει τη δυνατότητα να, να συνάπτει συμβάσεις. Από ό,τι βλέπω από την πρόταση θα διατηρήσει αυτό το δικαίωμα η Κομισιόν. Πρέπει να εξετάσουμε όμως προσεκτικά αν αυτός είναι ο κατάλληλος τρόπος για την οργάνωση του προγράμματος γιατί με τον τρόπο αυτό θα δημιουργήσουμε μια δεύτερη στρώση διαχειριστών και διαχείριση προγραμμάτων και μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση στο πρόγραμμα αυτό. Θα χαιρόμουν πολύ να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό στι επικείμενε διαπραγματεύσει. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Τσάνστονόφσκι. Συγγνώμη. Η κυρία Άντερς Δότερ πρώτα, ως πράσινη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας διαβεβαιώ ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα να με συγχαίρετε με τον κύριο Τσαρνόφσκι στην Επιτροπή αυτή. Θα ήθελα να τονίσω ότι είμαι διαθέσιμη να συνεργαστώ με τον εισηγητή και με τους άλλους κοιόδης εισηγητές για το θέμα αυτό. Είμαι πεπισμένη ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόταση αυτή είναι ενθαρρυντική. Η συνεργασία και η διαφάνεια είναι θετικά πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μας δίνει <clears throat> μεγαλύτερη δύναμη. Είναι πολύ καλό το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπογραμμίσει την ανάγκη συνεργασία και διαφάνεια. Το γεγονό ότι παρουσιάζει λύσεις η Κομισιόν για την πρόσβαση στα δεδομένα και την ιδιοκτησία των δεδομένων, αυτό είναι θετικό, πρέπει να εξετάσουμε όμως και τις λεπτομέρειες. Εγώ πιστεύω πρέπει να υπάρξει ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα και ελεύθερη ροή πληροφοριών. Το να εκχωρήσουμε στην Κομισιόν όμως το δικαίωμα να καθορίσει ποιος, έχει και ποιος, όχι, ποιος δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα, είναι κάτι που δεν με βρίσκει σύμφωνη, γιατί εγώ θέλω να προωθήσουμε την καινοτομία, να έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβαση για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και θέλω να παίξει μεγαλύτερο ρόλο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο ΕΣΑ, η οποία ήδη λειτουργεί σαν ένα φορέα συνεργασία, βοηθάει πολλά κράτη-μέλη και εγώ ελπίζω λοιπόν ότι θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου θα έχουμε περισσότερα, data, περισσότερα δεδομένα data σε όλους και θα μπορέσουν αυτό να είναι η βάση της συνεργασίας μας για το μέλλον. Ευχαριστώ. Τώρα ο κ. Τσαρτζενόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για το έργο του κυρίου Πρόντι, για την έκθεσή του, διότι πραγματικά έχει δουλέψει σκληρά και να μην επαναλάβω όσα υπόθηκαν. Συμφωνώ με το μεγαλύτερο μέρος. Όμως, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι το Κοπέρνικους, ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά απλώ άλλαξε όνομα, δεν θα πρέπει να επαναλάβει όσα γίνονται ως προς τις δράσεις και τη χρηματοδότηση αυτά τα στοιχεία, από τα στοιχεία άλλων προγραμμάτων. Εάν λοιπόν δεν απλουστεύσουμε την γραφειοκρατία, θα είναι σαν ε, να επαναλαμβάνουμε άλλα προγράμματα στα πλαίσια και του Κοπέρνικου. Θα πρέπει τα δεδομένα να διατίθενται με έναν τρόπο απλό, να υπάρχουν σαφή κίνητρα, είτε πρόκειται για δεδομένα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικού σκοπού, είτε άλλο τύπου, και να είναι απλή η πρόσβαση. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε νέου φορεί, οργανισμού ή συμβούλια διαχείρισης ή συμβούλια, τα οποία μπορεί στη συνέχεια να παρουσιάσουν προβλήματα ως προς την συνοχή τους. Θα πρέπει απλώς να έχουμε συνέστηση και συνείδηση ότι υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός του Διαστήματος και έτσι δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε κάποιες δραστηριότητε, ούτε τη χρηματοδότηση, αλλά ούτε και τις γραφειοκρατικές προβλέψεις. Πολλά υπόθηκαν ήδη, δεν θέλω να μακρηγορήσω, περνάει και ώρα, απλώς να πω ότι με μεγάλη χαρά θα συμμετάσχω στην περαιτέρω εξέταση του θέματος με τον κύριο Πρόντι, εκ μέρους ε, των Ευρωπαίων Μεταρρυθμιστών και Συντηρητικών. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα αυτό και θα πρέπει να έχουμε μια σαφή προσέγγιση. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Τσεφρανόφσκι. Όπως είπαμε, η έκθεση αυτή υπόκειται στους κανόνες του άρθρου 40, οπότε έχουμε υπεύθυνη εισηγητρία και από την ε, Επιτροπή Προπολογισμών, η οποία είναι και μέλο αυτή τη Επιτροπή. Κυρία Καρβάλιο, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Πρόντι, καθώ και εγώ ως σκιώδης εξήγητρια να πω ότι συμφωνώ με όσα ακούστηκαν, να κάνω μόνο μερικά σχόλια για το σκέλος του προϋπολογισμού. Από την πλευρά του προυπολογισμου οπως όπως ξέρετε, υπάρχει ειδική γραμμή 1α ε, με 3,76 εκατομμύρια για το 2011. Η δημοσιονομική γραμμή αυτή εγκρίθηκε και στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, οπότε θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το πρόγραμμα αυτό για να λειτουργήσει έχει επαρκή χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να προστατεύσουμε και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο προπολογισμός είναι πλέον σταθερός. Απλώς στη γνωμοδότησή μας σημαίνουμε ότι οι πρόσθετες ε, επιπλέον οικονομικές υποχρεώσεις θα πρέπει να ανακτηθούν μεταξύ των οροφών του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και του, των ίδιων πόρων. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος χωρίς να αντλήσουμε από άλλα προγράμματα όπως το Horizon 2020, το Γαλιλαίο και ούτω καθεξής. Άλλα που υπόκειται στο 1α. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Επιτροπή Προπολογισμών. Και το αναφέρουμε και στην γνωμοδότησή μας. Ένα δεύτερο σχόλιο στα πλαίσια των όσων είπαν και οι συνάδελφοι για την ε, διακυβέρνηση, τη διαχείριση του προγράμματος δηλαδή. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η διαχείριση αυτή είναι κάπως ασαφής. Θέλουμε κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο. Ε, θέλουμε να υπάρχει ένα πρότυπο διαχείρισης πιο ε, αναλυτικό και περισσότερες πληροφορίες προς το Ευρωκοινοβούλιο θέλουμε. Θα πρέπει να διδραματίζει έναν ενεργότερο ρόλο το Ευρωκοινοβούλιο στην παρακολούθηση της εξέλιξης του προγράμματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης θα πρέπει εγκαίρως να προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με το πρόγραμμα ως προς τη διαχείριση, το χρονοδιάγραμμα και τις επιδόσεις του. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Καβάλιο, ο κύριος Γκλάντε έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο λόγια μόνο. Καταρχάς ευχαριστώ τον συνάδελφο Ρωμάνο Πρόνταλο, του είπα και κάτι Ναι, συγγνώμη <laughs> Βιτόριο, με συγχωρείς, με συγχωρείς, με συγχωρείς. Κάποτε όμως κάποιος ε, υπήρξε, δεν υπήρξε Ρωμάνο. Λοιπόν, το θέμα της πολιτικής ε, για τα δεδομένα ε, μας είχε απασχολήσει και με τη σχετική οδηγία για την ελεύθερη και ανοιχτή πρόσβαση, free and open access. Τώρα λοιπόν μας έρχεται με διαφορετικές προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λεφτά όμω προέρχονται από την τσέπη του Ευρωπαίου φορολογουμένου. Δεν μπορεί να ε, χρησιμοποιούνται για σκοπούς που επιβαρύνουν τον φορολογουμένο. Πρέπει να βρούμε όμω κάποια λύση με υφιστάμενα επιχειρησιακά πρότυπα να δώσουμε λύσει, ε, ώστε να μην χρειαστεί να αντλήσουμε από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, παραδείγματι. Και ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, ναι, διμερείς με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ καλά. Αλλά να δούμε και τι δεδομένα μας δίνουν. Αν μας δίνουν δωρεάν ε, δεδομένα με ευκρίνεια 20 ε, μέτρων, ίσως είναι σκόπιμο να δούμε και σε απόσταση ενός μέτρου, η ευκρίνεια ενός μέτρου, πόσο μας ζητούν να πληρώσουμε. Ίσως ε, υπάρχει ζήτημα σε σχέση με, τις, ε, ε, με τα στοιχεία τα οποία αντλεί κανείς από το ραντάρ και αν αξίζει τον κόπο να εγκαταστήσουμε με δεδομένα αυτά ολόκληρο σταθμό στο διάστημα. Μήπως πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό και κατά πόσο αξιοποιείται ο Κοπέρνικος κατά τρόπο οικονομικό. Όλα αυτά λοιπόν και βέβαια στο βαθμό που μας αρκεί ο προϋπολογισμός είναι χρήσιμο, πολύ να τα ξανακοιτάξουμε. Ίσως Υπάρχουν κάποια όμως προβλήματα προς τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ κύριε Κλάντε. Η Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστώ τον κύριο Πρόντι για την έκθεσή του. έχει καλύψει πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα που πρέπει να κοιτάξουμε. Έχει αξιοποιήσει διατάξεις της οδηγίας Genesis και νομίζω ότι αυτό αποτελεί καλό ιονό και προοπτική για συμφωνίες από το Συμβουλίο. Ελπίζω δε ότι και τα δύο θεσμικά όργανα θα συμφωνήσουν συμφωνούν αρκετοί ότι υπάρχει πρόβλημα στον προπολογισμό, ότι έχει μειωθεί σε σχέση με τις αρχικές ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, η χρηματοδότηση. Φυσικά και δεν μας ικανοποιεί αυτή η κατάσταση. Συζητήσαμε το θέμα με την ε, ίσα και είπαμε ότι υπάρχει δυνατότητα για αναβολή των δραστηριοτήτων. Η ίσα μπορεί να προσφέρει 1,6 δις ευρώ ε, ώστε να καλύψει μέρος να δαπανών για την εκτέλεση του προγράμματος και έτσι μπορούμε με αυτές τις δύο συνδυασμένες ε, προτάσεις να χρηματοδοτήσουμε το συνολικό πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν. Τώρα, εάν καθυστερούμε λίγο στην προσοχή γενναία, θα έλεγα δεκαετία περισσότερο, σε αυτό οφείλεται. Η πολιτική και τα δεδομένα η αρχή της αμοιβαιότητας από ό,τι βλέπω είναι αυτή που υποστηρίζουν οι περισσότεροι ομιλητές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υποστηρίζει τη λύση αυτή, διότι η αμοιβαιότητα είναι προς όφελος μίας μόνο χώρας της Κίνας, η οποία είναι η μόνη χώρα που έχει ή θα έχει συγκριτικό, ε, μια συγκριτική σειρά δορυφόρων με αποτέλεσμα τα κινέζικα δεδομένα, να κατακλείσουν τις ευρωπαϊκές αγορές και ως εκ τούτου θα είναι ακόμα πιο περιορισμένες δυνατότητες αγοράς δεδομένων από εμά, αφού θα είναι δωρεάν όλα αυτά τα κινέζικα δεδομένα διαθέσιμα. Επίσης, σημειώνω τόσο είπε ο κ. Γκλάντ ε, για τη σχέση με τις ΗΠΑ καθώς οι ΗΠΑ έχουν αποστείλει δωρεάν δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δεκαετίες χωρίς επιβάρυνση. και θα πρέπει να συστήσουμε σοβαρά το τι είδου ε, δεδομένα θα αποστέλουμε και πώς θα τα χρεώνουμε. Αλλά όπως είπε ο κ. Γκλάντ, πρέπει να είναι συγκρίσιμη η ευκρίνη, η ποιότητα των δεδομένων. Και πριν καταλήξουμε σε συμφωνία για οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών, δεδομένων με τις ΗΠΑ, θα πρέπει να συμφωνήσουμε στο θέμα αυτό. Τη συγκρισιμότητα δηλαδή της ποιότητας των ε, δεδομένων. Εφόσον εξασφαλιστεί αυτό, θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή. Ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους διότι πέρασαν στην ουσία και τις έχουν μελετήσει τις προτάσεις μου με μεγάλη προσοχή. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα αισιόδοξο, διότι πιστεύω θα καταφέρουμε να ε, καταλήξουμε σε συμφωνίες λόγω και της πίεσης χρόνου, με την πίεση του χρόνου μάλλον ως δεδομένο, για να έχουμε ένα ε, καλό κείμενο. Να επιμείνω στο ότι το Κοπέρνικους ως διάδοχο πρόγραμμα του GMAS είναι άκρο σημαντικό. Εγώ είχα ενδιαφερθεί για το διάστημα από παλιότερα. Δεν είχα ενδιαφερθεί μάλλον για το διάστημα νωρίτερα. Όμως ε, το πρόβλημα που έθεσε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και τέθηκε εκεί πώς να καταμετρήσουμε λόγω χάρη τον άνθρακα που μπορεί να δεσμεύσει ένα δάσος το οποίο παρακολουθείτε και προστατεύεται, αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που μπορεί να το κάνει το GMAS, όπως μπορεί να κάνει και το Κοπέρνικος. Επίστηκα λοιπόν ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο και θα γίνει είτε για την διαχείριση του προγράμματος ανταλλαγής εκπομπών, του συστήματος μάλλον ανταλλαγή δικαιωμάτων εκπομπών, είτε για τα δεδομένα καταμέτρησης της υπερθερμάνσης του πλανήτη. Και προκειμένου να είμαστε σε επιφυλακή και να παρακολουθούμε τα των κλιματικών αλλαγών. Είναι άκρος απαραίτητο το εργαλείο αυτό να διατεθεί ως το δυνατόν συντομότερα στους χρήστες του. Και μάλιστα σε όλους τους ενδιαφερόμενους ε, χρήστες με την αμεβαιότητα που έλεγα. Δεν μιλάμε για αμεβαιότητα ταυτόχρονη. Θα μπορούσε λόγω χάρη. Και κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, που δεν έχουν ε, κάποιον ε, συνομιλητή να μας δώσουν δεδομένα. Είναι και θέμα καλής αγωγής να συμπεριφερέται έτσι κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με κάποια σχετική ταχύτητα προκειμένου να μπορέσει η εξέταση του θέματος να ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της θητείας μας. Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο διότι το Κοπέρνικος είναι εργαλείο απαραίτητο. Πρέπει λοιπόν να το έχουν στα χέρια τους αυτοί που το χρειάζονται. Όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η προθεσμία για τροπολογίες είναι η 3η 27 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Εντάξει, τελείωσε η συνεδρίασή μας. Η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 4 Νοεμβρίου στις 3 ώρα το απόγευμα και μετά στις 5 Νοεμβρίου το πρωί στις 9 εδώ στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και παρακαλώ να μείνουν οι συντονιστές τώρα για το, τη συνεδρία των συντονιστών. Περιμένουμε. everyone who's not allowed to be in here.